Λοιπόν, τα μέτρα ασφαλεία του Κοινοβουλίου τώρα επέτρεψαν πλέον στον Επίτροπο Αλμούνια να έρθει στην αίθουσα και τον καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μα. Στι 22 Μαρτίου ήταν η τελευταία φορά που είχαμε ανταλλαγή απόψεων ε, και στι 22 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και την επόμενη φορά τη συζήτησή μα. Δεν ξέρω γιατί τυχαίνει πάντα 22 του μηνό. Πάντως σήμερα δεν είναι στις 22 Ιουλίου. Θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο για 10 περίπου λεπτά και θα συνεχίσουμε στη, με τη συνήθεια ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχει η έκθεση της Επιτροπής ε, για τον Ανταγωνισμό το 2010 ε, που εκδόθηκε στις 20 Ιουνίου νομίζω και δεν είχαμε την ευκαιρία να τη συζητήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και τα θέματα ε, ενίσχυση για την κρίση. Αλλά θα υπάρχουν και άλλε ερωτήσει από του βουλευτέ. Υπάρχουν ε, τρία θέματα στον τομέα του ανταγωνισμού αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για αυτά τα θέματα μετά την παρουσίασή σα. Έχουμε την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεταρρύθμιση ε, των κρατικών ενισχύσεων για τι υπηρεσίε γενικού ε, συμφέροντος και τις συλλογικές προσφυγές. Αυτά είναι τα τρία θέματα που θα συζητήσουμε ως εκθέσεις ε, μετά τη δική σας παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Πάντοτε για μένα είναι μεγάλη χαρά να συμμετέχω σε ανταλλαγέ απόψεων με την Επιτροπή για Εικόν. Ευχαριστώ την Πρόεδρο Σάρων Μπόουλ για την ε, πρόσκλησή τη να περιβρεθώ εδώ. Και όπω ήδη είπε, το βασικό μου θέμα σήμερα θα είναι η έκθεσή μα για την πολιτική ανταγωνισμού το 2010. Και θα ήθελα να πω επίσης ε, δύο λόγια για το ψήφισμά σας μετά την έκθεση της πολιτικής ανταγωνισμού το 2009. Στο τέλος της σύντομης παρουσίασής μου, επειδή παρουσιάζουμε νέους κανόνες ανταγωνισμού για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που στο τέλος του έτους θα είναι έτοιμα, θα σας ενημερώσω για τη διαδικασία μεταρρύθμισης αυτών των ενισχύσεων. Έχουμε φέτος τη 14η έκδοση της Τη συγγνώμη, 400η έκθεση της ε, πολιτικής ανταγωνισμού. Είναι μια διαδικασία που έχει αναγνωριστεί ε, στο πέρασμα των ετών και βέβαια με ε, τα στοιχεία τα οποία εμείς ε, εκδίδουμε και με τον έλεγχο του ανταγωνισμού πολλοί είναι δυσαρεστημένοι αλλά μακροπρόθεσμα νομίζω ότι είναι προς όφελος όλων. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για το διάλογο σε αυτό το τομέα και για την υποστήριξή σας για τους στόχους της πολιτικής ανταγωνισμού. Όπως γνωρίζετε, το έργο για τις πολιτικές ανταγωνισμού κατά το περασμένο έτος ήταν ιδιαίτερα εντατικό. Εισαγάγαμε νέους κανόνες για την αγορά και για τις οριζόντιες και κάθετες συμφωνίες και ξεκινήσαμε μια σταδιακή έξοδο από το καθεστώς των ενισχύσεων για την κρίση ε, και ασχοληθήκαμε επίσης ε, και με τον χρηματοπιστωτικό τομέα λάβαμε πολλές αποφάσεις για τον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, όχι μόνο για τι τράπεζε, Πάνω από 400 αποφάσεις ελήφθησαν ε, υπό το φυσιολογικό καθεστώς. Επίσης, ε, πέρυσι ε, λάβαμε 14 αποφάσεις κατά των συμπράξεων και συμφωνιών ε, ήδη, ίδια επίπεδα ρεκόρ όπως το 2007 και 2008 και για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις επίσης είχαμε έντονη δραστηριότητα μετά τις επιπτώσεις της κρίσης τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι λάβαμε 270 κοινοποιήσεις και φέτος φαντάζομαι θα έχουμε και περισσότερες. Στι 7 αποφάσει για τις συμπράξει που λάβαμε πέρυσι επιβάλαμε πρόστιμα 3 εκατομμυρίων ε, ευρώ σε 17 εταιρείε και μειώσαμε τα πρόστιμα για 9 από τις 17 εταιρείε για να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των εταιριών σε οικονομικές δυσκολίες ε, στον, στην αντιμονοπολιακή νομοθεσία θα μιλήσω για το τομέα ενέργειας, μεταφορών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στον τομέα των μεταφορών η ε, απόφαση μας ε, αφορά τις ε, αεροπορικές εταιρείες ούτως ώστε να είναι προς όφελος των καταναλωτών τα μέτρα και οι αποφάσεις θα επηρεάσουν θετικά 2,5 εκατομμύρια επιβάτες. Στον τομέα της ενέργειας μετά την έρευνα που κάναμε το 2007 λάβαμε τέσσερις αποφάσεις σχετικά με τις εγκατεστημένες εταιρείε Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία για να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό στην αγορά. Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα ήθελα να επαναλάβω ε, τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Visa για ε, τα τέλη τα οποία επιβάλλει και αυτό αποτελεί ένα βήμα προόδου προς ένα σύστημα πιο αποτελεσματικό στον τομέα των πληρωμών ε, στην εσωτερική αγορά. Ξέρω ότι συζητάτε ένα αντίστοιχο θέμα αυτήν την εβδομάδα με την ψηφοφορία σας για, για τη ΣΕΠΑ, για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Πληρωμών. Εξετάζουμε επίσης τις πρακτικές των μεγάλων χρηματοπιστωτικών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών ω τμήμα τη πρώτη μα έρευνα στον τομέα των παραγόγων αυτές οι έρευνες δίνουν το μήνυμα ότι η κατάχρηση της αγοράς δεν θα γίνει ανεκτή και ότι η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα στον κανονισμό. Όλες αυτές οι αποφάσεις ε, θα βελτιώσουν τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη που είναι ένας κέριος στόχος ε, αυτός καθεαυτός. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς έχει και στρατηγικές επιπτώσεις και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναντι των διεθνών μας εταίρων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ενιαία αγορά εάν δεν μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς προβλήματα και η ενέργεια και τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν θέλουμε ε, να άρουμε τα εμπόδια τα οποία εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, δεν θα είμαστε σε θέση να προωθήσουμε τα οικονομικά μας συμφέροντα και τις αξίες μας στην διεθνή αγορά, στη διεθνή σκηνή. Τώρα θα ήθελα ε, να μιλήσω για τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμά σα για την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού τη Επιτροπή το 2009. Καταρχήν θέλω να επενέσω την εξαιρετική εργασία του εισηγητού σα, κυρίου Έπινγκ, και θα έχετε ήδη λάβει την επιστολή μου που απαντά όλα τα θέματα τα οποία συστήγεται στο ψήφισμά σα. Θα ήθελα απλώ να προσθέσω σύντομα σχόλια για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ε, για την επιβολή τη νομοθεσία στην αντιμονοπολιακή νομοθεσία και στι μελέτε που ζητήσατε να διεξαγάγουμε. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι μια μείζον πηγή απασχόληση, ανάπτυξη και καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντοτε αποτελούν τον πυρήνα των αποφάσεών μας για την επιβολή της νομοθεσίας. Βεβαίως θα διασφαλίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι, θα είναι συμβατές με, με την πολιτική ανταγωνισμού όπως και οι μεγαλύτερες εταιρείε, αλλά παράλληλα προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το διοικητικό άχθος που επιβάλλουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι νομοθεσίες μας. Θα σας δώσω λίγα από τα παραδείγματα των προσπαθειών μας. Στις κρατικές ενισχύσεις έχουμε τον κανονισμό για τις απαλλαγές κατά κατηγορία στον τομέα αντιμονοπολιακής νομοθεσίας νομοθεσίας, ε, ε, ε, η νομοθεσία de minimis εξαιρεί από τον έλεγχό μας τη συμφωνία μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μικρά μερίδια αγορά. και τέλο υπάρχουν νέοι κανόνε για να διευκολύνουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μικρομεσαίε επιχειρήσει. Παραδείγματο χάρη έχουμε τι οδηγίε για τα κεφάλαια κινδύνου. Επιπλέον, τα αιτήματα για μείωση των προστήμων λόγω τη μη δυνατότητα πληρωμής αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια τη κρίση και πέντε από τι εννέα εταιρείε που έλαβαν μείωση το 2010 ήταν μικρομεσαίε επιχειρήσει. Εξετάζω αυτή τη στιγμή πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας εταιρείε που κυρίως είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, όταν έχουν ε, ένα προϊόν και μόνο και αυτό να λαμβάνεται υπόψη όταν ε, επιβάλλουμε πρόστιμα για να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Το ψήφισμά σας επίσης εξετάζει την ανάγκη νομοθεσίας για να διευκολύνουμε την, τον αποτελεσματικό, την αποτελεσματική αντιστάθμιση για ζημίε που προκύπτουν από παραβίαση του αντιμονοπωλιακού δικαίου. Και συμφωνώ με όλα αυτά. Οι επιχειρήσει και οι καταναλωτέ στην Ευρώπη, ιδίω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και οι καταναλωτέ, θα πρέπει να έχουν την αντιστάθμιση στην οποία έχουν δικαίωμα. Και όταν μιλάμε για αντιστάθμιση και αποζημίωση για προσωπικέ ζημίες, έχουμε κατά νου και τι συλλογικέ προσφυγέ για τι οποίε ξεκινήσαμε διαβούλευση μέσα σε αυτή τη χρονιά. Λάβαμε με πάνω από 300 απαντήσεις μεταξύ αυτών και από πέντε αρχές ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε λάβει πάνω από 18.000 επιστολές από πολλούς ε, πολίτες. Είναι μεγάλη αριθμή αυτή και δείχνουν ότι και οι φορείς αλλά και οι απλοί πολίτε είναι έτοιμοι για μια πολιτική συζήτηση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα τεθούν επιτάπητο σε σημαντικά ζητήματα. Τώρα που ολοκληρώθηκε η διαβούλευση, προγραμματίζει η Επιτροπή μια ανακοίνωση για τις γενικέ αρχέ τη λογικής προσφυγή μέχρι τα τέλη του έτου. Και όταν οριστούν πλέον αυτέ οι αρχέ θα συζητήσουμε το πώς θα συνεχίσουμε τη δράση μας και στο δικό μου τομέα πώς θα συνεχίσουμε τη δράση μας ε, ούτως ώστε να επιβληθεί η νομοθεσία ε, στην πράξη. Τέλος, σας περάσουμε στις μελέτες. Η έρευνα που ζητήθηκε από το ψήφισμά σας αφορούσε κυρίως μια ανάλυση των επιπτώσεων των προσωρινών κανόνων κρατικών ενισχύσεων τους οποίους επιβάλαμε για να βοηθήσουμε το χρηματοπιστωτικό τομέα στην εποχή της κρίσης. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε λίγες εβδομάδες και τα αποτελέσματά της θα σας αποσταλούν και θα ανακοινωθούν πλήρως πλήρως ε, μετά το τέλος των διακοπών. Επίσης ε, είδα τη μελέτη που ζήτησε το Κοινοβούλιο για το ίδιο θέμα και χαίρομαι που μπορώ να παρατηρήσω ότι η έκθεση αυτή, παρότι είναι λιγότερο εκτεταμένη από τη δική μας έκθεση, κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα. Παραδείγματο χάρη και οι δύο μελέτες διαπιστώνουν ότι οι ενισχύσει που δίδονται στο χρηματοπιστωτικό τομέα είναι αιτιολογημένες και βοήθησαν να σταθεροποιηθεί η χρηματοπιστωτική αγορά και να παραμείνουν οι ε, ροέ προ την πραγματική οικονομία. Επίση, οι μελέτε παρατηρούν ότι η ε, χορηγηθή ενίσχυση δεν επηρέασε την ανταγωνιστική δομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τραπεζικό τομέα στο σύνολό του. Ωστόσο, η δική σα ε, μελέτη παραγνωρίζει ένα σημαντικό τμήμα της δράσης μας κατά τη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή τις διαρθρωτικές συνθήκες και την αναδιάρθρωση που επιβάλαμε στους κύριου αποδέκτε κρατικών ενισχύσεων. Η μελέτη μα δίνει λεπτομερεί πληροφορίε για αυτήν την αναδιάρθρωση που βασίστηκε σε προ... προσεκτικέ εξετάσει των περιπτώσεων στι οποίε βασίσαμε τι αποφάσει μα. Οι διαδικασίε αναδιάρθρωση που επιβάλλαμε σε ευρωπαϊκέ τράπεζε ελαχιστοποιούν τι τρευλώσει ανταγωνισμού που θα είχαν προκληθεί από τι ενισχύσει και εξασφαλίζουν την κατανομή βαρών μεταξύ των εμπλεκομένων. Τέλος, το πεδίο ε, εφαρμογή τη έκθεσής μας είναι ευρύτατο και έχει λάβει υπόψη του όλα τα θέματα. Λόγω ε, του εύρου της έκθεσης μπορέσαμε να καλύψουμε και άλλα θέματα όπως είναι η συνεισφορά των κρατικών ενισχύσεων σε μια πιο πράσινη ανάκαμψη. Πριν κλείσω την παρέμβασή μου, θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα το οποίο θα συζητήσετε αυτή την εβδομάδα, τη μεταρρύθμιση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για τι επιχειρήσει γενικού οικονομικού συμφέροντο. Ε, μετά την τελευταία ανταλλαγή απόψεων που είχαμε το Μάρτιο, συναντήθηκα με, την, ε, με τον κλάδο, με τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εταιρείε δημόσιε και ιδιωτικέ ε, που διεξάγουν δραστηριότητε γενικού οικονομικού συμφέροντο και με εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών. Ο διάλογος αυτός έχει δώσει χρήσιμα στοιχεία για τη σύνταξη των νέων ε, κανόνων μας και προετοιμάζουμε τρία εργαλεία τα οποία θα καλύπτουν τους βασικούς τομείς της μεταρρύθμισης. Μία ανακοίνωση η οποία θα διευκρινίσει τις βασικές έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να ασκήσουμε τον έλεγχό μας και που δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν οι εμπλεκόμενοι ε, όπως, όπως έχει τώρα. Δεύτερον, μια απόφαση που θα χρησιμοποιηθεί για να εφαρμόσουμε μια πιο απλή και πιο ευέλικτη προσέγγιση για τις τοπικές υπηρεσίες και ορισμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Και τέλος, ένα πλαίσιο που θα λάβει υπόψη του μεγάλα ποσά συμψηφισμού που χορηγούνται σε φορείς εκτός των κοινωνικών υπηρεσιών. Να σας πω ποιες είναι οι βασικές καινοτομίες αυτού του νέου πακέτου. Καταρχήν, θα ε, παρουσιάσουμε ένα κανόνα de minimis που θα είναι συγκεκριμένο για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος που θα, από όπου θα αποκλείονται ε, τα πολύ μικρά ποσά συμψηφισμού. Και για να υπάρχει πραγματικά τοπικό χαρακτήρα των υπηρεσιών που παρέχονται, αυτό ο κανόνα ε, θα εξαρτάται και από άλλα, κριτήρια, όπω το μικρό μέγεθο ε, των τοπικών αρχών αυτοδιοίκησης, το μικρό μέγεθο ε, των παρόχων υπηρεσιών. Δεύτερον, θα επεκτείνουμε το εύρο των κοινωνικών υπηρεσιών που εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίηση προ το, το παρόν καλύπτει μόνο νοσοκομεία και κοινωνική στέγαση. Τέλο, προτείνω η μελέτη μα να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίε θα παρέχονται γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά. Σύμφωνα με την παρούσα δέσμη μέτρων, η αποζημίωση που χορηγείται για την παροχή υπηρεσιών μπορεί να καλύπτει όλα τα στοιχεία κόστου ε, του παρόχου συν ένα λογικό περιθώριο κέρδου. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στοιχεία κόστου που αντισταθμίζονται από τα κρατημέλη μπορεί να οφείλονται σε χαμηλά επίπεδα αποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών και αυτό μπορεί να στρεβλώνει τη λειτουργία των αγορών και να πλήττει την ποιότητα των υπηρεσιών. Όσον αφορά τη διαδικασία, η μεταρρύθμιση βρίσκεται στο τελικό τη στάδιο. Τα κείμενα θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και θα δημοσιευθούν για δημόσια διαβούλευση τα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα συζητηθούν με τα κράτη-μέλη τον Οκτώβριο και αν όλα πάνε κατευχήν, οι νέοι κανόνε θα υιοθετηθούν κατά τα τέλη Ιανουαρίου του 2012. Βεβαίω με μεγάλη μου χαρά θα συζητήσω το θέμα αυτό μαζί σα και πάλι το φθινόπωρο πριν από την ε, τελική υιοθέτηση αυτή τη δέσμη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε. Να περάσουμε απευθείας στις ερωταπαντήσεις. Έχουμε περίπου μια μισή ώρα, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ακούμε μια φορά, κάθε φορά μάλλον από έναν συνάδελφο. Και για την ώρα έχουμε τον κύριο Σφάπ, την κυρία Πόδηματά, τον κύριο Κόπελτ, την κυρία Ίντφελτ, τον κύριο Σάντσες Πρεζέντο, τον Πίτερ Σίμον, την Αλίσσα Φερέρο, Φερέρα και τον κύριο Χοκμάκ. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Ωραία. Ανδρέας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω την υπηρεσία ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τη συγχαρώ για την εργασία στον τελευταίο καιρό Αυτό αυτά που αναφέρονται στην έκθεσή σας είναι μια εργασία που δεν είναι σημαντική όχι μόνο για την οικονομική κρίση, αλλά πολύ πιο γενικά. Και τονίσατε ότι η συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Γενοβουλίου εδώ και 40 χρόνια λειτουργεί ευτυχώ στον τομέα τη πολιτική του ανταγωνισμού. Και γι' αυτό θα θέλαμε επίση να σα ευχαριστήσουμε για την τόσο καλή και επιτυχή συνεργασία, ιδίω όσον αφορά την ανταλλαγή των απαραίτητων πληροφοριών. Ορισμένοι τομεί του οποίου τονίζει η έκθεση αναγνωρισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτο, τα τονίζατε. Θα ήθελα να, τονίσω, να προσθέσω κάποιου τομεί που νομίζω θα άξιζε επίση να αναφερθούν. Καταρχήν, θα ήθελα να τονίσω ότι όσον αφορά τα χρηματικά πρόστιμα στο τομέα του ανταγωνισμού και αυτό που αναφέρεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κατά πόσο δηλαδή οι υπολογισμοί βάσει των κατευθυντήριων ε, γραμμών βασίζονται στην απαραίτητη νομική βάση μακροπρόθεσμα ή κατά πόσο θα πρέπει να εξετάσουμε του κανόνε υπολογισμού και τι αρχέ επιβολή των προστήμων και αν θα πρέπει να ενταχθούν στον κανονισμό 1-2003 και αυτό το αναφέρατε τα, οι λεγόμενες υπηρεσίε ενός προϊόντος, ε, μόνο product businesses. Δεύτερον, και στον τομέα της ενέργειας όπου έχει δοθεί, που έχει δοθεί τώρα στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού από την ε, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, ΤΡΑΝ, υπήρξαν κάποιες αλλαγές τα τελευταία χρόνια ιδίω όσον αφορά ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2010, όπου μας δίνει τη δυνατότητα την εσωτερική αγορά ενέργειας και την απαραίτητη επιβολή και εφαρμογή της δέσμης των μέτρων για την εσωτερική πολιτική ενέργειας, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά, αλλά πρέπει ακόμα περισσότερα να κάνουμε. Τέλος, όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία, ο στόχος σας η πολιτική μας αναγωνισμού να είναι δηλαδή επιτυχής μακροπρόθεσμα μόνο αν ενταχθεί σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο είναι απόλυτα σωστή. Και θα ήθελα να τονίσω ένα σημείο. Στην Ελβετία, μια χώρα που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, εξακολουθούν οι υπηρεσίες αναγωνισμού αυτής της χώρας να μην είναι πλεγμένες να το πω έτσι στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο θα έπρεπε και όσο θα δικαιολογεί το λόγο των συνόρων που έχουμε τόσο πολύ με την Ελβετία. Τέλος, όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, θα επανέλθουμε αργότερα, αλλά ήθελα εδώ να τονίσω ότι κατά τη γνώμη μου η πρόταση που υποβάλλατε καλύπτει σε πολλά σημεία τα συμφέροντα των άμεσα ενδιαφερομένων. Και γι' αυτό η αναγγελία σας το φθινόπωρο να υποβάλλει μια νομοθετική δέσμη και για το θέμα αυτό ε, θα πρέπει να αναφερθεί η δέσμη για τα μέτρα του κοσμού. Κατά τα άλλα, χαίρομαι για την αλλαγή απόψεων και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση μέχρι το τέλειο. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Σφαμπ για το θέμα των προστήμων, χρηματικών προστήμων. Θεωρώ ότι η νομική μας βάση είναι πολύ σταθερή. Μπορείτε να δείτε και την νομολογία του δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο, όπου συμφωνεί πλήρως με τη δική μας νομική ερμηνεία πριν την ε, επιβολή ποινών ή συγκεκριμένα χρηματικών προστήμων. Αυτά βασίζονται στην ε, συνθήκη, στις αρμοδιότητες που αναθέτει η συνθήκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελευταία φορά το 2006 είχαμε ετοιμάσει για τα πρόστιμα κατευθυντήριες γραμμές, τις υλοποιούμε και Πρόσφατα λάβαμε τις πρώτες αποφάσεις του δικαστηρίου που αφορούν αποφάσεις οι οποίες απορρέουν από τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές. Νομίζω ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου επιβεβαιώνουν τις μεθόδους που ακολουθούμε. Συγκεκριμένα υπάρχει θέμα για ένα συγκεκριμένο πρόστιμο, όχι όμω για την νομική βάση, αλλά για τον τρόπο που εφαρμόστηκε. Πάντω, όπω είπα και στην παρουσίασή μου, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το πώ να απαλείψουμε ή τέλο πάντων να περιορίσουμε τη διακριτική μεταχείριση που σε κάποιε περιπτώσει παρεμποδίζει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει από το να είναι παραγωγικές. Σας το είπα και στην πρώτη μας συνάντηση, στην προηγούμενη συνάντηση, ότι έχω σκοπό να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, έχοντας ε, και πλέον ενό έτους πείρα επιβολής των ε, νέων μέτρων για, την, για τα χρηματικά πρόστιμα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό αυτό το συγκεκριμένο θέμα να εξεταστεί. Ίσως σε μια από τις επόμενες αποφάσεις μας για τα καρτέλ και τους ομίλους να μπορέσουμε να επανεξετάσουμε την αποφασή μας αυτή. Για την ε, ενέργεια, σας είπα ότι το θεωρούμε αυτό πολύ σημαντικό και ως προς τις κρατικές βοήθειες και ως προς τα τράστ που μπορεί να δημιουργηθούν. Συνεχίζουμε λοιπόν τις εργασίες μας σχετικά ε, και δεν πάβει να αποτελεί αυτό προτεραιότητα και ως προς τα μέτρα που θέλουμε και ως προς το οικοδόμημα που θέλουμε να φτιάξουμε και για την αγορά και για την ε, ε, εφαρμογή τη στρατηγική μα για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές. Η πολιτική ανταγωνισμού εδώ είναι ένα πανίσχυρο ε, όπλο και θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε. Κατανοώ τι ανησυχίε σα για κάποιες χώρες που δεν είναι ακόμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον βρίσκονται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ακολουθούν την ίδια γραμμή με εμά σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της πολιτικής ανταγωνισμού. Εργαζόμαστε εντατικά στο διεθνές προσκήνιο, ώστε οι διεθνείς αρχές ανταγωνισμού να συμμετέχουν. Ε, πρόσφατα συναντηθήκαμε στην ετήσια συνάντησή μας στη Χάγη και εκεί υπήρχαν ομάδες εργασίας, ομάδες δράσης. Συζητήσαμε διαμακρών με τις διάφορες εθνικές αρχές ανταγωνισμού και ελπίζουμε ότι η Ελβετία και άλλες τρίτες χώρες προοδευτικά θα συγκλίνουμε το δικό μας ε, πρότυπο, τις δικές μας μάλλον αρχές. Ε, στην ουσία εκπροσωπούμε οικουμενικότερες αρχές ανταγωνισμού που νομίζω ότι μπορούμε να τις ακολουθήσουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Ποδηματά στη συνέχεια. Και μετά ο Φιλίπ έχει ζητήσει το λόγο νωρίτερα από την προέβλεπη σειρά του, γιατί θέλει να πάει να ψηφίσει σε μια άλλη επιτροπή. Εάν κάποιος άλλος έχει παρόμοιο πρόβλημα χρόνου να μας το πει. Κύριε Αποκνοτά. Thank Ευχαριστώ. Σάρων, ευχαριστώ Επίτροπε για την παρέμβασή σας. Θα ήθελα να αποφεληθώ της παρουσίας σας εδώ, πριν ακριβώς από τις καλοκαιρινές διακοπές, διότι έχουμε πάλι μια κρίση σε σχέση με το δημόσιο χρέο στην Ευρωζώνη. Ένα θέμα που σχετίζεται λοιπόν με το χαρτοφυλάκιό σα και που εσεί έχετε θίξει σε διαφορετικέ περιστάσει. Ποιο είναι ο ρόλο των οργανισμών αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα. Από τη δική του πλευρά δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνουν υπόψη του κανόνε περί ανταγωνισμού. Αυτό το έχετε αναφέρει κι εσεί σε πολλέ διαφορετικέ περιπτώσει. Υπάρχει άλλωστε πολύ αρνητικό αντίκτυπο από τη λειτουργία τους, από τη βαθμολόγηση που επιβάλλουν και στο πώς εξελίσσεται η κρίση της Ευρωζώνης. Επιτροπή, η ερώτηση μου είναι η εξή. Η Επιτροπή θα αντιδράσει για το θέμα αυτό πριν είναι πλέον πολύ αργά. Εδώ και εβδομάδες, εδώ και μήνες παρακολουθούμε αυτό το περίεργο, το παρά, την παράξενη ανάμιξη των οργανισμών αυτών στις ε, συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των διαφόρων θεσμικών φορέων όμως. Θεσμικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε σχέση με το τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει το νέο πακέτο υποστήριξης για την Ελλάδα συγκεκριμένα. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι το δικό του το πόρισμα η δική τους η αξιολόγηση καθορίζει το αν θα υπάρξει περίπτωση στάσης ή αν θα υπάρξει ένα πιστοτικό γεγονός. Εκείνοι φαίνεται να δίνουν την τελευταία λέξη για το όλο πρόγραμμα ε, ή για το αν θα υπάρξει ανάμειξη του ιδιωτικού φορέα στην ε, επίλυση της κρίσης. Ε, ξανά λοιπόν θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν η κρίση επεκταθεί και γίνει ένα φαινόμενο ακόμη πιο επικίνδυνο, πιο γενικευμένο που θα πλήξει ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ποια είναι η δική σας η άποψη. Τι λέτε για τις ιδέες που ακούστηκαν στο να δημιουργηθεί πλέον ένας ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Ε, και τέλος, πώς αντιδράτε σε αυτό που είπε ο Επίτροπος πριν από λίγες μέρες, ότι η βαθμολογία από αυτούς τους η βαθμολογία των κρατών μελών από αυτού του οργανισμού και μάλιστα η βαθμολογία κρατών που ήδη βρίσκονται σε ένα πρόγραμμα προσαρμογή δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Τι άποψη έχετε για αυτή τη δήλωση, Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ. Κατά πρώτον, είναι πολλέ οι φωνέ που ακούγονται, ιδίω τι τελευταίε εβδομάδε και ημέρε, και αναφέρουν δημοσίω ότι οι οργανισμοί εξόλευση πιστολιτικής ικανότητας είναι ο λιγοπόλιος στην ουσία. Και ισχύει αυτό γιατί έχουμε μόνο τρεις τέτοιους οργανισμούς. Ευθύ αμέσω λοιπόν αντέδρασα ενημερώνοντα τη δική μα ανάλυση, ζητώντα τέλο πάντων από τι υπηρεσίε μου να επικυροποιήσουν την ανάλυση τη όλη κατάσταση από την σκοπιά τη πολιτική ανταγωνισμού. Πρέπει να πω ότι από αυτήν ακριβώς τη σκοπιά πρέπει να δούμε τις περιπτώσεις κατάχρησης ε, επικρατούσας θέσης, ή τις ε, δράσεις που μπορεί να προκύπτουν από το άρθρο 1.1 της συνθήκης. και που μπορεί να έχουν σχέση με τις δραστηριότητες αυτών των οργανισμών. Πάντως πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τις δυνατότητες αντίδραση σε σχέση με αυτά τα λιγοπόλια και το τι αντιμετώπιση μπορεί να έχουμε μέσω, από την, μέσω της πολιτικής ανταγωνισμού. Αυτό είναι κάτι που καθημερινά με απασχολεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαστόματος του Επιτρόπου κ. Μπαρνιέ και του Πρόεδρου τη του κ. Μπαρόζο ανακοίνωσε ότι ετοιμάζουμε ένα νέο κανονισμό για αυτού του οργανισμού. Τον τρίτο κατά σειρά από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Θα συζητηθεί το θέμα και θα εκφράσω και εγώ τις απόψεις μου σε αυτή τη συζήτηση στο κολέγιο. Δεν θα το συζητήσω δημοσίως πριν ληφθεί μια απόφαση σε επίπεδο κολεγίου επιτρόπων, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσον υπάρχει και η πιθανότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Ε, μπορώ να σας πω τις δικές μου τις απόψεις για το θέμα αυτό. Δημοσίως ακόμη όχι, αλλά πρέπει να κάνω τα εξή τρία σχόλια. Πρώτα απ' όλα είναι προφανές ότι ο ρόλος των οργανισμών αυτών από την αρχή αυτής της κρίσης ήταν πολύ κακός, απέσιος εξ αρχή συμπεριφέρονται με πολύ λανθασμένο τρόπο. Η δική του αξιοπιστία είναι πλέον πολύ χαμηλή. Η αξιοπιστία τους ήταν ε, ιδίω πολύ χαμηλή στην αρχή τη κρίση, όταν ανέλησαν τους κινδύνου και έδωσαν βαθμούς ε, για τα ενεργητικά του ιδιωτικού τομέα. Τώρα νομίζω ότι πραγματικά χάνουν ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία τους και από την πλευρά του δημοσίου τομέα. Όμως δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε την αξιοπιστία. Δεν είναι αντικειμενικό στοιχείο αυτό, αλλά νομίζω ότι πραγματικά η αξιοπιστία του αυτή τη στιγμή όλο ένα και υπονομεύεται, μειώνεται. Ας είμαστε όμω σαφείς για να επιλύσουμε τα προβλήματα κάποιων ε, οικονομιών της Ευρωζώνης. Και οι παρελκόμενε συνέπειε που δημιουργούν για την υπόλοιπη περιοχή σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικέ αποφάσει. Εγώ θεωρώ ότι η δική μου η ευθύνη, όπως και των υπόλοιπων ηθινόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρώ ότι οι υποφάσεις αυτές επήγουν. Δεν μπορούμε πλέον να αποποιούμαστε των ευθυνών μας, να αναλάβουμε, να λάβουμε αποφάσεις και να τα ρίχνουμε όλα στις οργανισμούς. Ευχαριστώ, Φίλιπ. Ευχαριστώ, Σάρων. Έχω δύο ερωτήσει, ε, κύριε Επιτροπέ. Η μία αφορά μία από τι πρόσφατε ε, δηλώσει. Εκεί που λέτε ότι τελευταία καναλή κλείδι υπάρχουν πάρα πολλέ τράπεζε στην Ευρώπη, θα ήταν καλύτερα να, έχετε, να έχουμε λιγότερε και πιο μεγάλε. Μου φαίνεται περίεργο ένας ε, επίτροπος υπεύθυνο για τον αγωνισμό να λέει κάτι τέτοιο. Γιατί θέλετε από την άλλη μεριά η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική με τους διεθνείς μας εταίρους θα πρέπει να έχουμε αρκετά μεγάλες βέβαια επιχειρήσεις. Από την άλλη μεριά ο τραπεζικός τομέας ε, νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από τράπεζες υπορβικά μεγάλες και έχουμε πολλές. Θα έπρεπε να μειώσουμε το μείδος ορισμένων γιγάντων του τομέα. που στρεβλώνουν την αγορά κατά βάση και όχι να τονίζουμε το γεγονό ότι υπάρχουν πολλέ μικρέ τράπεζε που ορισμένες από αυτέ μάλιστα δεν έχουν τόσο καλή διαχείριση. Και μετά θα ήθελα να υποβάλω την ερώτηση που υπέβαλα και πέρσι. Ανησυχώ ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού δεν ενδιαφέρεται για τον ε, διακριτικό χαρακτήρα που δίνει η Κεντρική Τράπεζα στον τραπεζικό τομέα. Γιατί η Κεντρική Τράπεζα κρατά στη ζωή ορισμένε τράπεζες που άμα τι είχαμε αφήσει στη μοίρα τους θα είχαν πτωχεύσει. Και αυτέ είναι τράπεζε που δεν τυχάνουν καλή διαχείριση. Γιατί εκείνε που τυχάνουν καλή διαχείριση δεν έχουν ανάγκη από τι ενίσχυσει τη κεντρική τράπεζα. Έχουμε λοιπόν εδώ μια έντονη στρέβληση του ανταγωνισμού και δεν ξέρω ένα επικεφαλή του ανταγωνισμού θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Απάντηση του Επιτρόπου. Όσον αφορά τον αριθμό των τραπεζών, καμιά φορά με επικρίνουν γιατί η πολιτική μας ανταγωνισμού και οι αποφάσεις του Επιτρόπου για τον ανταγωνισμό είναι κατά της ύπραξης Ευρωπαίων πρωταθλητών και για να είμαστε ανταγωνιστικοί αν δούμε τι κάνουν οι ανταγωνιστές μας αλλού. Ακόμα και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένες χώρες. Υπάρχουν άλλες χώρες, άλλες αγορές που είναι εθνικές αγορές για τις τράπεζες που έχουν ελληνική αν θέλετε προσφορά, υποθήκη, δάνεια υποθηκών κλπ που δεν μπορούν να προχωρήσουν. Και ακριβώς το πολύ μικρό μέγεθος πολλών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι προβληματικό. Γιατί ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτεί την οικονομία μας. Είναι απαραίτητο. Η πολιτική ανταγωνισμού λοιπόν δεν έχει σαν στόχο να υποδιαιρεί το μέγεθος των επιχειρήσεων. Άλλος είναι ο στόχος της. Να αποφευχθεί η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης. Αλλά αν υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση που είναι ανταγωνιστική και από την άλλη μεριά σέβεται τους κανόνες της αγοράς και δεν οδηγεί σε στρέβλωση της αγοράς, θαυμάσια. Για τους καταναλωτές που θα πρέπει να είναι εκείνοι που θα ωφεληθούν από την πολιτική ανταγωνισμού. Λοιπόν, Επιμένω σε αυτή τη δήλωση. Υπάρχουν ορισμένε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπάρχει πολύ μικρό αριθμό τραπεζών κατά τι κρίση. Το πιο ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ιρλανδία και στην Ιρλανδία έκανα κάποιες δηλώσεις πρόσφατα που είπα ότι θα πρέπει για να μειωθούν οι ησυχίε ε, στον οικονομικό τομέα, να δούμε τι θα γίνει με τον αναγνωρισμό στον τομέα αυτό το ίδιο ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο, που μειώθηκε ο αριθμό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην αγορά. Αλλά κοιτάξτε άλλε χώρε. Η δική μου χώρα τα ταμιευτήρια μειώθηκαν από 46 στα 15 στη χώρα μου και μου φαίνεται είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Δεν οδηγεί αυτό σε κινδύνους για τον ανταγωνισμό του αντίον, οδηγεί στην καλύτερη δυνατότητα αντιμετώπισης των ε, κινδύνων ε, της ε, προσοχής προς τους πελάτες κλπ όσον αφορά τις ενισχύσει της τράπεζας. Κατόπιν τη κρίση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, ξεκίνησε ένα καινούριο σύστημα ε, ενίσχυσης ορισμένων τραπεζών έναντι ε, στοιχείων, αν θέλετε, και πρέπει να τη συγχαρούμε γι' αυτό, γιατί αλλιώς πολλά από αυτά τα χρηματοπιστικά ιδρύματα, πολλές από αυτές τις τράπεζες δεν θα μπορούσαν να επιζήσουν. Αυτά τα μέτρα βέβαια δεν επιτρέπεται να διανυστούν. Εξορισμό. θα πρέπει σιγά σιγά να βγούμε από αυτού του τύπου το, το σύστημα. Τώρα το θέμα είναι ποιος πρέπει να βγει από το σύστημα και ποιος επιτρέπεται να συνεχίσει να λαμβάνει αυτή την έκτακτη βοήθεια και υποστήριξη. Για δείτε τι γίνεται στην Ιρλανδία για να ξαναπάρουμε το ίδιο παράδειγμα. Οι Ιρλανδικέ αρχές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να περάσουν σε μια διαρθρωτική βοήθεια και λέει η τράπεζα όχι, όχι και τη στηρίζω σε αυτό. Είναι μεταβατικά τα μέτρα αυτά, προσωρινά. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τις δικές μας απόψεις για την μεμονωμένη ευθύνη των Ιδρυμάτων δεν μπορούμε να κλείσουμε αμέσως αυτό το παραθυράκι ε, ρευστότητας. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της άγουσας. Προχωρήσαμε αρκετά, αλλά υπάρχουν και κάποια ακόμα οι ιδρύματα που δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς αναδιάρθρωση. Και κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης χρειάζονται εξαιρετική γραμμή αν θέλετε ρευστότητα από την Κεντρική Τράπεζα. Κάθε φορά που εξετάζουμε κάποια αναδιάρθρωση μεμονωμένη και έχουμε πάρει πάνω από 30 μεμονωμένες τέτοιες αποφάσεις και προετοιμάζουμε καμία κοσαριά άλλες και ίσως και άλλες αιτήσει να υποβληθούν. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι αναδιάστρωση, μείωση του συλλογισμού, ε, βιωσιμότητα του επιχειρησιακού μοντέλου, ε, των ε, εμποδίων ανταγωνισμού κλπ. κλπ. Αυτό κάνουμε εμείς. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων όμως να επικρίνουμε. Γιατί πρόκειται για μια μεταβατική αλλά απαραίτητη βοήθεια κατά τη γνώμη μας. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον Επίτροπο για την παρουσίασή του. Το διάβασα αναλυτικά στην έκθεσή του. Επιτρέψτε μου να υποβάλω μια ερώτηση. Η έκθεση συνοψίζει πάρα πολύ καλά τα διδάγματα στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε από αυτούς τους ελέγχους. Απ' την άλλη μεριά θεωρώ ότι η πολιτική ανταγωνισμού των τελευταίων ετών δεν άλλαξε όσον αφορά τις ευθύνες και τους επιμέρους τομείς. Αυτή τη στιγμή όμως η αλλαγή γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι χαρακτηριστικό για την σήμερα. Και στην έκθεση αυτή εγώ δεν βλέπω ποια είναι τα κίνητρα που θέλετε να δώσετε για το έτος 2010. Και πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτά. Σας παρακαλώ κύριε Επιτροπέ να μας παρουσιάσετε μια προφορική προσθήκη της έκθεσής σας. Και μια άλλη ερώτηση που αφορά επίσης τις τράπεζες. Αναφερθήκατε στις ενισχύσεις που είναι προσωπορινές και μεταβατικής μορφής μας είπατε. Επίσης Εάν κατάλαβα σωστά, είπατε ότι αυτό συνέβαλε στον ανταγωνισμό. Μα εγώ διάβασα κάποιες μελέτες οι οποίες ακριβώς ε, λένε το αντίθετο. Ότι η κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν βελτιώθηκε. Για στείλτε μας σας παρακαλώ μια, τη μελέτη αυτή στην οποία αναφερθήκατε που αποδεικνύει ότι βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητα. Δεν ακούστηκε πολύ καλά η πρώτη ερώτηση που μου κάνατε. Βλέπετε να υπάρχει κάποια έλλειψη στην έκθεση νομίζω, αλλά δεν κατάλαβα πού ακριβώς ε, πήγαινε αυτή η πρώτη ερώτηση, αν μπορούσατε να μου την επαναλάβετε. Δεύτερο ερώτημα. Για τις έκτακτες ε, βοήθειες προς την ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας και την ε, ανόρθωση του τραπεζικού τομέα. Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση του συστήματος που θα μπορούσε να παραλύσει τελείως τις οικονομικές ροές έπρεπε κάτι να γίνει και όταν προλάβει κανείς ένα τέτοιο κίνδυνο χάρη στην ε, ανόρθωση μπορεί να επιτρέψει να εργαστεί κανείς πλέον πάλι στην πραγματική οικονομία, στην Ευρώπη. και όσοι βασίζονται στις τραπεζικές, ε, εκείνοι μάλλον που βασίζονται στις τραπεζικές επιταγές κυρίως, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτοί η αλυσίδα πρέπει να ξαναλειτουργήσει με έναν τρόπο μάλιστα ευέλικτο και ώστε να μπορεί να δανειστούν χρήματα υπό τους σωστού όρου. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει οι οικογένειε να μπορέσουν να υποφεληθούν εφόσον το θέλουν. Να μπορούν να χρηματοδοτήσουν ε, τις αγορές τους, το ίδιο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι σαφές αυτό. Η μελέτη μα θα είναι έτοιμη στο τέλο του καλοκαιριού ή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει λοιπόν να αποτιμήσουμε τα όσα έχουν γίνει ως τώρα, να δούμε τι λύσεις υπάρχουν και να προχωρήσουμε τις προσπάθειές μας. Αυτό ακριβώς κάνουμε σε σχέση με την αναδιάρθρωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία και πάλι. Ελπίζω να μου επαναλάβετε την πρώτη σας ερώτηση που δεν κατάλαβα καλά. Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας κάνω ξανά την ερώτηση. Θεωρώ ότι υπάρχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στην έκθεση και βλέπω ότι ε, υπάρχουν πολλά στοιχεία και το θέμα που αφορά τα χρηματικά πρόστιμα επίσης. Αλλά όσον αφορά το 2010, με βάση τον προγραμματισμό σας, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να επιτύχετε. Είναι καλή η έκθεση, αλλά δεν έχω κάποιο επίπεδο αναφοράς. Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο είναι καλά τα αποτελέσματα και κατά πόσο χρειάζεται κάτι άλλο. Επίτροπος, ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω στην πρώτη ομιλία που είχα κάνει εδώ όταν ήμουν υποψήφιος επίτροπος τον Ιανουάριο του 2010. Ανέλαβα μια δέσμευση τότε, μιλώντας εκ μέρους ε, ολόκληρης της Επιτροπής, γιατί συζητούσαμε τις ε, πολιτικές ε, της Επιτροπής, αναλάβαμε μια δέσμευση συνολικά και πιο συγκεκριμένα για το πρώτο έτος της θητείας μας στην Επιτροπή. Αναλάβαμε κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες δεσμεύσεις και νομίζω ότι όλες οι δεσμεύσεις που ανέλαβα τότε κατά την ακρόασή μου τηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2010. Σόφη. Κυρία Ιντβέλτ. Α, συγγνώμη, δεν καταλάβα το όνομά μου. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πάντοτε χαιρόμαστε όταν έρχεστε εδώ. Έχω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, αναφερθήκατε στη Visa, τη Mastercard και τη συζήτηση που γίνεται ε, για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και θα ακούσατε και τα σχετικά με την ψηφοφορία ε, για το χώρο συναλλαγών ΣΕΠΑ. Συζητήσαμε λοιπόν αυτό το θέμα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ΜΙΦ. Νομίζετε ότι προχωρούμε αρκετά γρήγορα ώστε να διασφαλίσουμε επαρκή ανταγωνισμό και εύκολη πρόσβαση ε, σε νεοεισερχόμενους στην αγορά. Έχω την εντύπωση ότι αυτά προχωρούν πάρα πολύ αργά. Μια δεύτερη ερώτηση που έχει σχέση με τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Με ενδιαφέρουν πολύ οι προτάσεις σας και θα τις περιμένω. Παρ' όλα αυτά, είμαι κάπως δύσπιστη όσον αφορά τις γενικές εξαιρέσεις στις οποίες ήδη αναφερθήκατε. Αναφέρατε τα νοσοκομεία και είπατε ότι μπορεί να προκύψουν και άλλες κατηγορίες που θα εξαιρεθούν ως κατηγορία. Το πρόβλημα είναι ότι στα διάφορα κράτη-μέλη η διάρθρωση αυτών των θεμάτων είναι διαφορετική. Δηλαδή, ακόμη και τα νοσοκομεία σε ορισμένε χώρε μπορεί να είναι αντικείμενο εμπορική διαχείριση, σαν να ήταν μια εμπορική επιχείρηση. Γιατί να εξαιρούνται λοιπόν από του κανονικού κανόνε και να μην ε, υπόκειται στου γενικού κανόνε ανταγωνισμού. Οι γενικέ εξαιρέσει λοιπόν ε, ενέχουν κινδύνου και θα ήθελα η Επιτροπή να προσέξει πάρα πολύ στο τι κάνει σε αυτό το τομέα. Τρίτη ερώτηση. Είναι ερώτηση, αλλά δεν ξέρω βέβαια αν θα μου απαντήσετε. Στην έκθεσή μου για την πολιτική ανταγωνισμού, καθώς και αργότερα σε ανταλλαγές απόψεων στην ΕΚΟΝ, στην Επιτροπή μας, ε, ε, συνεχώς ε, συζητώ το θέμα της διαφήμισης στο διαδίκτυο και των μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο αν ξεκινήσει μια τέτοια έρευνα δεν θα μας το πείτε φαντάζομαι γιατί δεν θέλετε να πανικοβληθούν όλοι αλλά πριν από δύο εβδομάδες ακούσαμε ότι έχει ξεκινήσει μια βάση δεδομένων που ονομάζεται εξάξεις που περιλαμβάνει 500 εκατομμύρια ατομικά προφίλ κυρίως Ευρωπαίων πολιτών και υπάρχουν τόσο πολλές πληροφορίες για τους πολίτες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταγωνιστεί κανείς μια τέτοια προσπάθεια. Ξέρω ότι είναι νέος τομέας, είναι πιο εύκολο να εξετάσει κανείς τον τομέα της, παρα... παραγωγής προϊόντων όταν έχουμε απτά προϊόντα, αλλά στον τομέα του διαδικτύου έχουμε ένα τομέα με τεράστια ανάπτυξη και αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ινβέλτ. Πρώτον, όσον αφορά ε, ε, τα μυθ και τις ε, κάρτες που αναφέρατε, όπως επίσης και τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες. Εξετάζουμε τα θέματα αυτών των μυθ για τις πιστοτικές και κάρτες άμεσης χρέωσης και έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία με τη Visa που ανέλαβε δεσμεύσεις όπως και, για, όπως και η Mastercard αλλά για την άμεση χρέωση, όχι για τις πιστοτικές κάρτες. Αυτό είναι ένα θέμα που το εξετάζουμε ακόμη. Υπάρχουν κάποιοι ενδεχόμενοι εισερχόμενοι στην αγορά καρτών στην Ευρώπη και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε τις τράπεζες αυτές προς ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών με κάρτα. Κατά τη γνώμη μου, σε ορισμένα θέματα, ε, η άποψή μου λέω, είναι ότι θέλουν να είναι καλοί Ευρωπαίοι αλλά με υψηλό τίμημα και έχω κάποιες αμφιβολίες κατά πόσο θα επωφεληθούν δηλαδή οι Ευρωπαίοι καταναλωτές από μια ευρωπαϊκή κάρτα που θα είναι πιο ακριβή από τις άλλες. Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν. Και υπάρχει άλλη μια συζήτηση για τις κάρτες άμεσης χρέωσης και για αυτές ε, τις υπηρεσίες ε, πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες. και συζητάμε με τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις. Ε, το ερώτημά μου είναι, είστε σίγουροι ότι δεν χρειάζεται κάποια ρύθμιση του τομέα και έχουμε μια task force με τις υπηρεσίες του Μισελ Μπαγνιέ και με υπηρεσίες ε, της Γενικής Διεύθυνσης Υπεύθυνης για τους Καταναλωτές ακριβώς για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και για να το πω με διπλωματικό τρόπο, δεν το βλέπω τόσο εύκολο το να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα που έχουν σχέση με τα συστήματα πληρωμών και να ανοίξουμε τους φραγμούς για τα νέα συστήματα πληρωμών, εναλλακτικά συστήματα πληρωμών, χωρίς ρύθμιση το βρίσκω πολύ δύσκολο. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών το συντομότερο δυνατόν σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε αυτή την εσωτερική αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτό που είπα και στην απάντησή μου προ τον κύριο Λαμπέρ, τα χρειαζόμαστε αυτά και δεν είμαστε αρκετά ισχυροί για να επιλύσουμε τα προβλήματα και να άρουμε τους φραγμούς μόνο με εργαλεία ανταγωνισμού. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να έχουμε και ρυθμιστικά μέτρα. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή. Συμφωνώ μαζί σας λοιπόν ότι καθυστερούμε. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ στα βήματά μας προς ένα πραγματικό ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών ΣΕΠΑ. Συζητάμε και μπορούμε να συζητήσουμε και ενημερώσει αυτό το θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών και το, της ειδική μεταχείρισης. Οι περισσότερες από αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες και δεν είναι εύκολο να ορίσουμε το τι ακριβώς είναι κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών. Είναι πολύ λεπτή η διαχωριστική γραμμή. Αυτό θα καλύπτεται από την ειδική μεταχείριση για τις μικρές υπηρεσίες που παρέχονται, από τοπικές κοινότητες, ε, χωρίς να έχουμε στρεβλώσει ανταγωνισμού διαμεθοριακά κλπ. Πάντως εξαίρεση σημαίνει εξαίρεση από την, προηγούμενη, από την υποχρέωση προηγούμενη. Δηλαδή μιλάμε για κρατικές ενισχύσεις, υπάρχουν δηλαδή κρατικές ενισχύσεις, αλλά στις περισσότερες από αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες μπορούμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, πιστεύω, αν τους χορηγήσουμε εξαίρεση από την υποχρέωση κοινοποίησης και μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτεπαγγέλτος μία έρευνα και να ασχοληθούμε με τις καταγγελίες ή να εξετάσουμε τον έλεγχο εκ των υστέρων και να δούμε αν υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις για να έχουμε παραβίαση της νομοθεσίας. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει εξαίρεση. Για μένα εξαίρεση αφορά αυτό, αυτούς που είναι κάτω από το επίπεδο του de minimis και είναι πολύ μικρές αυτές οι εξαιρέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις στις κρατικές ενισχύσεις έχουμε υποθέσεις που απαιτούν πολλή δουλειά πρέπει να παρακολουθούμε δηλαδή τα όσα γίνονται και τελικά είναι πολύ μικρή η επίπτωση, είναι σχεδόν μηδενική η επίπτωση τη τρέβλωση ανταγωνισμού. Ε, Επομένω, ίσω είναι καλύτερα να αφιερώσουμε πόρου στι πραγματικά σημαντικέ περιπτώσει, παρά να κάτσουμε να ασχολούμεθα με λεπτομέρεια, με όλε τι περιπτώσει που πρέπει να αναλύσουμε και καταναλώνουν πόρου λόγω καταγγελιών που γίνονται και κοινοποιήσεων κλπ. Γι' αυτό είπαμε ότι μπορεί να έχουμε αυτή την εξαίρεση από την πρώτερη κοινοποίηση. Τώρα, για τι μηχανέ αναζήτηση και τι διαφημίσει ε, στο διαδίκτυο Αρχίσαμε τις έρευνες με το, για το Google πέρυσι. Το Google έχει το 94% της αγοράς μηχανών αναζήτησης σε αυτή την αγορά. Έχουμε πολλά λοιπόν να, δούμε και, έχουμε, και μαθαίνουμε πολλά. Δεν θα σας αποκαλύψω τώρα τα, τις λεπτομέρειες αυτής της έρευνας. Εξετάζουμε πιθανώς την πιθανή ύπαρξη στρέβλωσης ανταγωνισμού στις μηχανές αναζήτησης και όσον αφορά τον τομέα της διαφήμισης γιατί και οι διαφημίσεις είναι μια πηγή εσόδων για την Google. Μαθαίνουμε λοιπόν πάρα πολλά με αυτή την έρευνα που κάνουμε και για τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο, διαφημίσεις online. Αυτό δεν είναι αποκλειστική δραστηριότητα της Google. Ίσως λοιπόν από την υπόθεση της Google μάθουμε πάρα πολλά που θα μας βοηθήσουν και για άλλες περιπτώσεις. Νομίζω ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτό το τομέα είναι να προχωρήσουμε την έρευνά μας σε αυτό που κάνουμε με την Google δηλαδή αυτή τη στιγμή γιατί μαθαίνουμε πάρα πολλά όπως σας είπα πολύ ανησυχητικό είναι το ποιο έχει τα προσωπικά μα δεδομένα και πώ τα χρησιμοποιεί. Μιλάμε για την εφημερίδα News of the World τι τελευταίε ε, μέρε ε, και τα θέματα του ιδιωτικού απορρίτου είναι πολύ σημαντικά, αλλά είναι θέματα ιδιωτικού απορρίτου και όχι ανταγωνισμού αυτά τα θέματα. Αν γίνεται κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, μπορεί κανείς να επωφεληθεί και από την κατοχή προσωπικών δεδομένων που έχει. Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Κάποιοι φορείς της χρηματοπιστωτικής αγοράς εξετάζουμε πώς χρησιμοποίησαν τις πληροφορίες προς όφελός τους, πώς χρησιμοποίησαν την ισχύ που έχουν στην αγορά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση προσωπικών δεδομένων πρέπει να το εξετάσουμε. Αλλά καταρχήν πρόκειται για θέμα προστασίας δεδομένων και θέματα ιδιωτικού απορρίτου και το εξετάζει κατά αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή. Ίσως κάποια μέρα να ανοίξουμε την έρευνα και προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά μέχρι τώρα, όπως σας είπα, ασχολούμεθα με την έρευνα που αφορά την Google, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η έρευνα. Είναι μια βασική έρευνα που δεν είναι εύκολη γιατί είναι καινούρια και όχι μόνο καινούρια, αλλά είναι και ένας κινούμενος στόχος. Αυτός ο τομέας, αυτοί οι φορείς αλλάζουν συνεχώς τμήμα του επιχειρηματικού, του επιχειρηματικού τους μοντέλου και των βασικών τους δραστηριοτήτων τροποποιούνται συνεχώς. Άρα πρέπει και εμείς να ακολουθούμε αυτόν τον κινούμενο στόχο και αλλάζουμε συνεχώς το πεδίο της ερευνάς μας. Ευχαριστώ πολύ. Άντελη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φέτος είναι μια σημαντική χρονιά γιατί γιορτάζουμε την 40η επέτειο της πολιτικής ανταγωνισμού, την 41η συγκεκριμένα. Μιλήσατε λοιπόν για την αντιμετώπιση της κρίσης και ήθελα να σχολιάσω το θέμα των βοηθειών που προσφέρθηκαν. Δεν θα πρέπει οι δικαιούχοι των ε, των στήριξη να βρεθούν σε πλεονεκτική σχέση σε σχέση με όσου δεν έλαβαν στήριξη. Πρέπει να δούμε τη θέση την ανταγωνιστική όσων δεν έκαναν χρήση λοιπόν ε, των βοηθειών και τι γίνεται με τη θέση των τραπεζών στις κρατικές βοήθειες. Τι γίνεται, με τις τι γίνεται με την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πώς μπορεί να καθοριστεί η θέση που φέρνει κάποιον πλεονεκτική θέση σε σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού. Τώρα για τις αγορές και την πρόσβαση στις υπηρεσίες. εδώ για την πρόσβαση στις υπηρεσίες πρέπει να δούμε ακριβώς ε, τι πληρώνει ο καθένας και βεβαίως ε, τι πρέπει να αναλογίσει τον κάθε πολίτη. Το στοιχείο λοιπόν ε, πρόσβαση στην αγορά των υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικό και έπειτα για τις συναλλαγές και τις προμήθειες των διτραπεζικών συναλλαγών. Μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Κάρτα. Εδώ θα ήθελα μια διευκρίνηση. Μιλήσαμε για την πολιτική ανταγωνισμού και την, το κατά πόσον θα τεθούν εδώ κάποια κριτήρια την, με τη διαδικασία της συναπόφασης και για το διεθνές προσκήνιο. Σε αυτή τη φάση οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν έρευνες για παρα... περι... περιπτώσεις όχι μόνο εντός ΗΠΑ, αλλά και εκτός την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω Ε, θα πρέπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να κάνουμε κάτι ανάλογο. Θα πρέπει και εμείς να ξεκινήσουμε διαδικασίες έρευνας για ορισμένες συμπεριφορές στην αγορά, και σε στενή συνεργασία με τις Αμερικανικές αρχές. Νομίζω ότι και αυτό είναι καθοριστική σημασία, ώστε να γίνει αποτελεσματική και δραστική παρέμβασή μας και σε αυτό το πεδίο. Και έπειτα η σχέτιση του ανταγωνισμού με την ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει κάποιους τομείς όπως η γεωργία και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις να τις ε, δούμε ώστε να υπάρξει και ανταγωνιστικότητα αλλά και στρέβλους του αγωνισμού στην αγορά ή ε, η περιαγωγή. Εδώ ποιος είναι ο ρόλος της ανταγωνιστικότητας είναι σημαντικό με τους ισχύοντες κανονισμούς. Τέτοιου είδου διευθετήσει λοιπόν θα πρέπει να γίνουν έχοντα υπόψη και την ανταγωνιστικότητα. Πρόεδρο, νομίζω ότι οι ερωτήσει αυτέ ήταν πέντε στην ουσία. Θα πρέπει νομίζω να, τις δούμε, να απαντώνουν δύο βουλευτέ κάθε φορά πλέον. Ευχαριστώ να... πολύ. Να τα πω στη γλώσσα μου για να προσπαθήσω να είμαι και πιο σύντομο για την πρώτη ερώτηση. Δεν νομίζω ότι η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ρευστότητα, γιατί εδώ μιλάμε για δάνεια. Δεν νομίζω ότι ε, θα πρέπει αυτό να αποτελέσει ε, αντικείμενο ε, κοινοποιήσεων για κρατικές ενισχύσεις και υπάρχουν και ειδικέ ενισχύσει ρευστότητα, αυτό είναι μια ειδική πιστοτική γραμμή που χορηγήθηκε στο σύστημα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό ξεπερνάει ε, το θέμα των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και περνάει από, το, από τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όταν υπάρχει ε, ε, κρατική ενίσχυση στον τομέα των ενισχύσεων ή των, των εγγύησεων, όταν, όταν χορηγούνται πιστώσεις από κάποιο κράτος, και εδώ φτάνουμε σε αυτά τα οποία αποφασίστηκαν το 2008-2009 κατά την περίοδο της κρίσης. Παράλληλα εξετάσαμε και την απαραίτητη αναδιάρθρωση. Σαν αντιστάθμισμα προς τις πιστώσεις ζητήθηκε και αναδιάρθρωση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν και την αναδιάρθρωση τώρα. Όσον αφορά ε, τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, είναι τεράστιο το θέμα αυτό και συμφωνώ ε, με το γενικό πνεύμα της ερώτησής σας. Θέλω όμως να τονίσω ότι η ρύθμιση ε, στα θέματα κρατικών ενισχύσεων για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος με βάση το άρθρο 156 της συνθήκης δεν είναι ρύθμιση για όλες τις ε, υπηρεσίες ε, γενικού οικονομικού συμφέροντος. Ε, για ορισμένα θέματα συζητάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραδείγματο χάρη για τις καθολικές υπηρεσίες. Και στη συνθήκη αναφέρεται ότι το αφήνουμε στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών όταν υπάρχουν καθολικές υπηρεσίες η απόφαση για την καθολική υπηρεσία πολλές φορές δεν λαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή είναι μια απόφαση που λαμβάνει το κράτος μέλος χρησιμοποιώντας τη διακριτική ευχαίρεια που έχει σε αυτό τον τομέα. Καταλαβαίνω λοιπόν την ερώτησή σας, αλλά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να ρυθμίσουμε τις κρατικές ενισχύσεις με βάση ε, την ε, απόφαση Μόντι Cruz όπως πολλές φορές έχω πει στην Επιτροπή μας η Επιτροπή στην Επιτροπή σας η Επιτροπή επεξεργάζεται όλα αυτά τα θέματα και στα τέλη του έτους ε, θα περάσουμε σε ανακοίνωση μέτρων σχετικά με τη συλλογική προσφυγή για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον κάθε τομέα. Μας ενδιαφέρει και πώς επηρεάζεται ο ανταγωνισμός από το θέμα της συλλογικής προσφυγής, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. σε διάλογο με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αφού εγκρίνουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής επί της αρχής, θα συζητηθούν όλα αυτά. Η νομοθεσία μας θα βασίζεται στη διαδικασία της συναπόφασης και θα χρησιμοποιήσουμε την απαραίτητη νομική βάση ούτως ώστε να έχουμε συναπόφαση. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολύ σημαντική η εθνική νομοθεσία και χρειαζόμαστε συνεργασία και με τρίτες χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες. Στις Ηνωμένε Πολιτείες Υπάρχουν ε, εταιρείε για τι οποίε είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα τη αντιμονοπολιακής νομοθεσία, και έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τους ομολόγου μα στις ΗΠΑ και με το Υπουργείο Δικαιοσύνη και με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ανταγωνισμού. Και μεταξύ των υπηρεσιών μας έχουμε ακόμη και καθημερινές συνομιλίες και ανταλλαγή πληροφοριών, όχι βέβαια απόρριτων πληροφοριών, και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης παραδείγματο χάρη έχουν ε, κάποιους περιορισμούς, ιδίως στον ποινικό τομέα, όχι στον τομέα του αστικού δικαίου, οπότε υπάρχουν και κάποια θέματα απορρίτου, αλλά υπάρχουν ε, υποθέσεις τις οποίες σχεδόν ταυτόχρονα συζητάμε και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μερικές φορές μου λένε άλλοι επίτροποι, όπως ο κ. Μπαχνιέ, ότι είναι πιο δύσκολο να συντονιμάσαι από ότι να συντονιστούμε με εκείνους. Γενικώ δηλαδή έχουμε πολύ καλές σχέσεις και δεν υπάρχουν ε, παράπονα. Ε, στο παρελθόν ενδεχομένως υπήρχαν δυσκολίες, τώρα όμως δεν υπάρχουν ε, κάποιες δυσκολίες που χρειάζεται να αναφέρουμε. Για τα θέματα της συλλογική προσφυγής Έχουμε πει ότι ε, θα αποφασίσουμε ε, αμερόληπτα για οποιαδήποτε περιοχή και αν πρόκειται, είτε ε, σε μεγάλες είτε σε μικρές χώρες, στο βορρά είτε στο νότο. Μια εξαίρεση είχαμε κάνει στο γαλακτοκομικό τομέα ήταν η μοναδική. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τις συμπράξει σε κανένα τομέα. Στις τηλεπικοινωνίες έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Έλλη και οι υπηρεσίες μας ε, βρίσκονται σε ε, διαρκή ε, συζήτηση και έχουν πολύ καλή συνεργασία. Ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος της ρύθμισης και ποιος είναι ο ρόλος του ανταγωνισμού και σε όλες τις περιπτώσεις και στις τηλεπικοινωνίες και στο στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και στην ε, διανομή του φάσματος η συνεργασία μας είναι εξαιρετική. Χρησιμοποιούμε δηλαδή με έξυπνο τρόπο τα εργαλεία που διαθέτουμε και στον τομέα της ρύθμισης και στον τομέα του ανταγωνισμού για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Διάφοροι ζήτησαν το λόγο, οπότε προσθέθηκαν στον κατάλογο των αγορητών. Θα προσθέσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις πολλές μαζί. Ε, μην ε, μπείτε σε ανταγωνισμό να ρωτήσετε περισσότερα από τον προηγούμενο, αν μπορείτε. Τώρα ο Πίτερ Σάιμον και η κυρία Φερέιρα. Και μετά ο κύριος ε, Χέκμαρ και ο κύριος Χοντής. Κλείνω τον κατάλογο με την κυρία Γκουλάρ και οποιοδήποτε σκέφτηκε να ζητήσει το λόγο ε, αργότερα έχει χάσει. Πίτερ. Θα ήθελα να δώσω το καλό παράδειγμα. Γιατί αν δεν άρχισε με πέντε ερωτήσει, εγώ θα έχω μόνο τρει. Ο επόμενο λοιπόν μία ερώτηση και θα προφτάσουμε. Εγώ ζητώ το λόγο ω εισηγητή της έκθεσης πρωτοβουλίας για τη μεταρρύθμιση των ε, διατάξεων για τις κοινοτικέ ανεχίσεις για τις ε, υπηρεσίες ε, γενικού οικονομικού συμφέροντος. Και θα ήθελα εδώ κύριε Αλμούνια να σας ευχαριστήσω που αναφερόσαστε σε αυτό το κείμενο. Ήδη η ανακοίνωση που υπήρχε καταδεικνύει πόσο σοβαρά λαμβάνει υπόψη το θέμα αυτό και πόσο έχετε λάβει υπόψη τις δικές μας παρατηρήσεις ήδη. Και από προσωπικές συζητήσεις μαζί σας στο Στρασβούργο ξέρω ότι θα τις λάβετε και αυτές που ακούτε σήμερα υπόψη. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω που προσανατολίζετε το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας, από ό,τι μου είπανε, στις διαδικασίες του Κοινοβουλίου. Γιατί το Κοινοβούλιο άρχισε κάπως αργά να ασχολείται. Παρ' όλα αυτά θέλετε οι παρατηρήσει μα να μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την λήψη αποφάσεων. Τρει ερωτήσει. Χαιρετίζω τις σκέψεις όσον αφορά μία προσέγγιση διαφοροποιημένη για τις κρατικές ενεργήσει. στις υπηρεσίε γενικού οικονομικού συμφέροντος να υπάρχει δηλαδή για τις εν λόγω επιχειρήσεις ένας κανόνας de minimis που λόγω του περιορισμένου τοπικού του χαρακτήρα θα έχουν σχετικά ελαχιστοποιημένες επιπτώσεις στην ευρύτερη αγορά. Αυτό βοηθάει πολλά κράτη-μέλη γιατί διευκολύνει τη ζωή σε πολλούς τομείς. Εναντιάζει προς τον άνθρωπο Ίνφελτ όμως, θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση όσον αφορά τον τομέα της ε, υποχρέωσης κοινοποίηση, εξαίρετα ξέρετε νοσοκομεία κλπ. δεν υπόκεινται. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, θα μπορούσε να φανταστεί κανένα ότι και άλλε κοινωνικέ υπηρεσίε μπορούν να εξελιχθούν. Παραδείγματο χάρη η φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων με ειδικέ ανάγκε και γενικά του τομέα τη υγεία. Μία ερώτηση αυτή. Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται σε κάτι που συζητήσαμε στο Στρασβούργο, το θέμα δηλαδή της αποτελεσματικότητας των ε, υπηρεσιών αυτών ε, γενικού οικονομικού συμφέροντος, στο τελευταίο σημείο της ανακοίνωσης του Μαρτίου. Κατανοώ ότι η Κομισιόν θέλει να λάβει υπόψη και κριτήρια αποτελεσματικότητας στις μελλοντικές ε, μελέτες και καταλαβαίνω ότι ο ε, φορολογούμενο είναι κάτι τέτοιο ευκταίο. Αλλά δεν βλέπω που υπάρχει η νομική βάση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι υπάρχουν τα κριτήρια αυτά Αλμάρκ όπου αλλάζει και η στάση, η θέση μάλλον από την οποία μπορεί να κρίνει η Κομισιόν. Και αν υπάρχουν δηλαδή τέσσερα κριτήρια Αλμάρκ που να τηρούνται, πώς θα ελέγξει η Κομισιόν. Και τέλος, από τη δημοκρατική ε, σκοπιά, εμεί είπαμε πάντα ότι βάσει το άρθρο 14 οι αρχές και οι όροι για τη λειτουργία των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ε, θα πρέπει να υιοθετηθούν βάσει ενός κανονισμού από το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Η Κομισιόν πέρα από το θέμα που συζητάμε σήμερα μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα υποβάλει μια σχετική πρόταση. Ελίσσα, ah, uh, uh, μήπως μπορείς να ρωτήσεις και εσύ τώρα. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Είχα μόνον δύο ερωτήσει να θέσω. Πρώτα απ' όλα για την αδυναμία των τραπεζών ή τέλο πάντων τη στήριξη που, προσφέραμε στι τράπεζε σε τέτοιε δύσκολε στιγμέ. Νομίζω σε περίοδου κρίση, παρεμβάσει ήταν ε, χαρακτήρο κατεπήγοντο. Όμω, μου φάνηκε να αντιλαμβάνομαι από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30 Μαρτίου να προτείνεται μετά τα τεστ ε, κοποσος των ε, τραπεζών να αναλάβουν οι επιμέρους χώρες τις διορθωτικές παρεμβάσεις που χρειάζονται ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις των τραπεζικών τους τομέων. Άρα έχει αναβληθεί για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το Σεπτέμβριο. Η ανάλογη δράση όμως δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε αυτά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, θα έχουμε εθνικέ αγορέ πλέον τελείω ξεχωριστέ σε περίοδο κρίση για την αντιμετώπιση μάλλον των προβλημάτων κρίση των τραπεζών. Αυτό το βρίσκω ανησυχητικό. Και το δεύτερο μου ερώτημα έχει να κάνει και με το ερώτημα τη κυρία Ποδηματά. Έχω ενδιασμούς και αμφιβολίε όταν μου λέτε ότι στην περίπτωση των οργανισμών αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας δεν μπορέσαμε να κατηχωρήσουμε την κατάχρηση της δεσπόσουσας θέσης, τους ε, φραγμούς που μπορεί να υπήρξαν στην πρόσβαση, τις συμφωνίες που μπορεί να επετέφθησαν. Εδώ υπάρχει μια σειρά παραγόντων και στοιχείων, ε, μια ε, συγκυρία που δείχνει ότι υπάρχει ολοϊκοπόλιο και στρεβλώνει την αγορά. Θα ήθελα λοιπόν, αν έχετε, να μου πείτε ημερομηνίε συγκεκριμένε που να προβλέπονται για μια νέα απόφαση του Συμβουλίου του Κολεγίου των Επιτρόπων κατά πρώτον και μετά κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρξει μια καινούργια πρωτοβουλία για τον έλεγχο των οργανισμών αξιολόγησης. Αυτό θα πρέπει να γίνει και σε συνεργασία με τι ε, Ηνωμένε Πολιτείε βεβαίω, αλλά οπωσδήποτε κάτι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κατεπήγον. Συμφωνώ απολύτω με αυτό που είπατε. Ε, εδώ απαιτούνται πολιτικέ αποφάσει. Δεν μπορούμε να είμαστε χωρί πολιτικέ αποφάσει και χωρί μια σοβαρή εξέταση των, ε, των ε, καταστρεπτικών για τον ανταγωνισμό αποτελεσμάτων που έχει δράσει των ε, οργανισμών αυτών στην αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κατά πρώτον για τον κύριο Σίμων για την εξαίρεση από τις ε, απαιτήσει κοινοποίηση. Βάσει του πακέτου μετρών που ισχύει από το 2005, η εξαίρεση αυτή αφορά την κοινωνική στέγαση και τα νοσοκομεία. Εγώ πρότεινα να διευρυνθεί η εξαίρεση και για άλλες υπηρεσίες. Μια σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες που ήδη έχουν αρχίσει να συζητούνται με τους ε, αρμόδιους εμπειρογνώμονες Εντό των υπηρεσιών της Επιτροπής αλλά και με διάφορους παραγόντες των ε, κοινωνικών μα εταίρων, των κοινωνικών μας συνομιλητών. Ήδη είχα κάποιες πρώτε επαφές και χθε και εδώ στο Κοινοβούλιο και έχουμε διεξαγάγει μια σειρά συζητήσεων για να δούμε ποιε κοινωνικέ υπηρεσίες γενικού συμφερόντο θα πρέπει να καλυφθούν εδώ. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι τομείς που να μην βρίσκουν όλους σύμφωνους αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε όταν προκύπτει θέμα για τον κάθε επιμέρους τομέα. Όπως είπα προηγουμένως και στην κυρία Ιντβελτ, Τώρα για την αποτελεσματικότητα της ανταγωνιστικότητας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με την νομική βάση. Όταν βλέπουμε μέτρα λιτότητας, δημοσιονομικές περικοπές και περικοπές στις δαπάνες, λογικό είναι μια εταιρεία που προσφέρει γενικώ ε, υπηρεσίες να υποβάλλεται στον έλεγχο μια αρχής. Θα πρέπει δηλαδή να μπορεί να ελεγχθεί η ανάληψη τέτοιων υπηρεσιών από ένα πάροχο και να μπορεί να ελεγχθεί το κατά πόσον από την άποψη του κόστου και τη ωφελία είναι σωστή η σχέση, είναι ισόρροπη. Θα πρέπει λοιπόν οι πολίτε που αποφελούνται τέτοιων υπηρεσιών να ωφελούνται πραγματικά. Εάν υπάρξουν εξοικονομήσεις πόρων, θα πρέπει το κέρδος να το μοιράζονται οι κοινωνικοί εταίροι και οι δημόσιες αρχές ενδεχομένως. Αυτός ο κανόνας ισχύει λόγω χάρη για τις ε, χερσαίες ε, συγκοινωνίες. Είναι λοιπόν νομίζω λογικό κάτι τέτοιο και επωφελές για όλους τους πολίτες. Δεν βλέπω να υπάρχει λοιπόν σχετικά πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι λογικό να περιμένουμε από κάποιον που παρέχει δημόσιες υπηρεσίες να εργάζεται πιο αποτελεσματικά. Και όσοι θα, θα λάβουν τα κέρδη από την αύξηση της αποδοτικότητας ε, ενό τέτοιου φορέα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τις δημόσιες αρχές. Τώρα, ο η νομική βάση για την εξέταση του θέματος αυτού είναι το άρθρο 106. Όπως απήντησα και στον κύριο Σάντσες Πρεσέντο προηγουμένως, υπάρχουν κάποιες ε, κάποιοι ενδιασμοί σε σχέση με το άρθρο 14, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων για την παροχή υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Εκεί όμως σίγουρα η νομική βάση είναι το 106. Το άρθρο 14 αναφέρει ότι με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων σε ό,τι αφορά τι κρατικέ ενισχύσει. όταν αναφερόμαστε σε άλλες πτυχέ των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντα. Όταν, ε, ε, αν στραφώ τώρα στην ερώτηση της κυρίας Φερέιρα, τα τεστ κοπόσεως για τις τράπεζες. Ήδη έχουν διεξαχθεί κάποια συμπεράσματα και ρωτήσαμε τα κάτι μελη το εξή. Είστε πρόθυμοι όταν δημοσιευθούν τα αποτελέσματα των τεστ κοπόσεως να τροφοδοτήσετε με πρόσθετα κεφάλαια ώστε να καλυφθούν οι απατούμενες υπηρεσίες και αυτό ήδη πολύ σύντομα ώστε να μην έχουμε προβλήματα στάσεων, πληρωμών ή στρεβλώσεων της αγοράς. Οι ανεπάρκειε του συστήματο ήταν κάτι που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε και στο παρελθόν κατά τη διάρκεια τη κρίση. Το Συμβούλιο, λοιπόν, κατά την άποψή μου, ορθώ είπε ότι πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε να αυξήσουμε τα κεφάλαια στι αγορέ. και αν οι αγορέ δεν είναι σε θέση να τροφοδοτήσουν με αρκετά κεφάλαια κάποιον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ένα αποθεματικό έτοιμο, αποθηκευμένο, ώστε να αξιοποιηθεί εκείνη τη στιγμή. Λέει ο κανονισμό ότι για κάθε ευρώ που δαπανάει η δημόσια αρχή σε κάθε χώρα, για, μια, για έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό, για να αυξήσει δηλαδή αυτός ο οργανισμός το κεφαλαίο του, ή για να εκδώσει ένα κρατικό ομόλογο, ή για να στηριχθεί σε σχέση με τα τοξικά τέλο πάντων παράγωγα, θα πρέπει για κάθε τέτοιο ευρώ ο χρηματοπιστωτικό οργανισμό να υποβάλει ένα σχέδιο αναδιάρθρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εμεί θα πρέπει να αξιολογήσουμε αυτό το σχέδιο αναδιάρθρωση. Την μείωση του ισολογισμού, των δαπανών στον, του παθητικού στον ισολογισμό, την, τα μέτρα αναδιάρθρωση, το πώ θα είναι βιώσιμο πλέον αυτό ο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Αυτό σημαίνει την ε, ε, σωστή ε, κατεύθυνση των επενδύσεων, την σωστή επιλογή επενδύσεων και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν κάθε στρέβλωση προ τον ανταγωνισμό λόγω τη κρατική ενίσχυση να απελευθεί. Μόλι λάβει κανεί ένα ευρώ κρατική ενίσχυση για την αναδιαρθρώση θα πρέπει να υποβάλει και το ανάλογο σχέδιο. Ήδη έχουμε λάβει 20 τέτοια σχέδια, τα εξετάζουμε και είμαι σίγουρο θα λάβουμε πολύ περισσότερα στο μέλλον. Τρει χώρε τη Ευρωζώνη βρίσκονται σε πρόγραμμα ε, δημοσιονομική αναδιάρθρωση. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία έχουμε δει τα προγράμματα της κάθε μιας χώρας ξεχωριστά. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε και άλλα σχέδια από άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο μέλλον και για τους οργανισμούς αξιολόγησης. δεν θα πάψω κάθε μέρα να θέτω το ερώτημα προς τις υπηρεσίες μου κατά πόσο να έχει υποβληθεί κάποια προσφυγή. Εάν υπάρξει παραμικρή προσφυγή για την κατάχρηση ε, της δεσπόζουσας θέσης στην παράβαση του άρθρου 101, ε, θα αναλυφθεί αμέσω δράση. Για την ώρα δεν υπάρχουν τέτοιε προσφυγέ, ούτε υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία στη σημερινή συγκυρία, ώστε να ξεκινήσει μια επίσημη έρευνα. Αυτό πάντω που υπάρχει είναι σαφώ μια δέσμευση τη Επιτροπή να υποβάλει ένα νέο σχέδιο κανονισμού το φθινόπωρο. Αυτή θα είναι η τρίτη πρωτοβουλία μα από τότε που ξεκίνησε η περίοδο τη κρίση και εγώ συμφωνώ ότι αυτή η ανάγκη είναι επιτακτική. Υπάρχουν διαφορετικέ μεν απόψει για το πώ να διευθετήσουμε την κατάσταση και το κατά πόσον μπορεί να χρειαστεί ένας ευρωπαϊκός ε, οργανισμός εδώ, όπω υπενήφθηκε και η κυρία Ποδηματά. Όμω, ε, εδώ για την αξιοπιστία των οργανισμών Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε εδώ ότι αυτή η αξιοπιστία σαφώς έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα τον τελευταίο καιρό. Το ακούσαμε ήδη. Ε, παραμένει όμως γεγονός ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας με το βαθμό που θα ανακοινώσει αμέσως επηρεάζει τις αγορές. Έχει άμεσο αντίκτυπο η δράση του. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την περασμένη μόλις εβδομάδα ε, έκανε νομίζω ένα πολύ σωστό βήμα σε σχέση με την περίπτωση της Πορτογαλίας. Είπε δεν με νοιάζει ποιος είναι ο βαθμός του οργανισμού του οποιοδήποτε. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο σε σχέση με το δημόσιο χρέο ε, και του οργανισμού. Ευχαριστούμε, Γκούναρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επανέρχομαι στο θέμα των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος που έχει συζητηθεί και από πολλούς προαναλύσαντες. Διαβάζοντας την ανακοίνωση αλλά και από τη συζήτηση αυτή βλέπω ότι κυρίως εστιάζονται τα θέματα στο πώς μπορούμε να διευκρινίσουμε, να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες και νομίζω ότι αυτό και σωστό είναι και σημαντικό και συμφωνώ απολύτως. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να προσθέσουμε άλλη μία οπτική γωνία, δηλαδή πρέπει να απλουστεύσουμε και να διευκρινίσουμε και το πώς μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη σε αυτούς τους τομείς. Και νομίζω ότι αυτή η πτυχή λείπει, για να είμαι ειλικρινής όσον αφορά την ανακοίνωση δεν υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση, δηλαδή ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει καλύτερη δυνατή εξέλιξη σε αυτούς τους τομείς, γιατί είναι τομείς πολύ σημαντικοί για τους πολίτες, για τα κράτη-μέλη και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αν δείτε κάποιες τέτοιες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, σαφώς είναι και κέρια σημασία για τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη, για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Και το ερώτημα είναι, ε, έχουμε ανταγωνιστικούς τομείς και έχουμε τον ανταγωνισμό που απαιτείται. Παράλληλα με αυτό πρέπει να ε, βοηθούμε τους παρόχους να εξελίσσονται. Αν δούμε το ιστορικό βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια αλλαγή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, παραδείγματο χάρη. Δεν θα θέλαμε να το έχουμε αυτό και στον τομέα των μεταφορών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών, της ενέργειας και σε άλλους τομείς. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση λείπει, κύριε Επίτροπε. Όταν θα έρθετε λοιπόν να μας υποβάλλετε την πρότασή σας, νομίζω ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια τέτοια πτυχή. Διότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ κρατικών ενισχύσεων προς τους παρόχους ή προς τις υπηρεσίες. Διαφέρουν οι παραδόσεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνετε την πρότασή σας με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν περισσότερες διασυνοριακές δραστηριότητες, να υπάρχουν περισσότεροι κορυφαίοι πάροχοι σε αυτούς τους τομείς όχι μόνο απλούστευση και διευκόλυνση δηλαδή, αλλά και κάτι παραπάνω. Διότι αν δεν υπάρχει η πιο δυναμική προσέγγιση της εξέλιξης, ο κίνδυνος είναι ότι απλουστεύουμε μόνο και μόνο για να διατηρήσουμε τις σημερινέ δομές που δεν είναι ανταγωνιστικές, που δεν συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα που χρειάζεται η Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω πώς θα χειριστείτε αυτό το θέμα. Πρέπει να τηρήσουμε την επικουρικότητα και τις διαφορετικές παραδόσεις των κρατών μελών, αλλά παράλληλα Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και νέοι πάροχοι υπηρεσιών, μεγαλύτερη πολυφωνία. Διαφορετικά αυτό θα αποτελέσει τροχοπέδι για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Επαναλαμβάνω λοιπόν όχι μόνο απλούστευση και διευκρίνηση αλλά και εξέλιξη της αγοράς. Ευχαριστώ. Νίκολας, ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αλμούνια, σας ε, ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ και επειδή σε λίγη ώρα θα τελειώσει η τελευταία συνάντησή μας πριν από τις διακοπές, σας εύχομαι καλές διακοπές. Αλλά σας παρακαλώ, για να μην με βασανίζουν ενδεχομένως και άλλους συναδέλφους κάποια ερωτήματα στις παραλίες, δώστε μου κάποιες απαντήσεις για να μπορέσουμε να περάσουμε ήσυχα. Πρώτο θέμα επανέρχομαι στο θέμα των οίκων αξιολόγηση, αξιολόγησης. Συγγνώμη, διότι είπα μια έκφραση που κολλάει πολύ για το χαρακτηρισμό. Ή και αξιολόγησης. Λοιπόν. Είπατε διάφορα. Διαβάζω σήμερα ο κύριος Μπαρνιέ, η κυρία Ρέντινγκ, πριν λίγες μέρες ο κύριο, κύριος Μπαρόζο, καταφέρεστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για τους οίκους αξιολόγησης. Και σας ρωτώ, είπατε ότι το φθινόπωρο σε ερώτηση συναδέλφου τιμάζεται τον τρίτο κανονισμό. Μπορείτε να μου πείτε ποιος τίμασε το δεύτερο κανονισμό και αναφέρομαι στα ονόματα γιατί είσαστε παλαιότερα μέλη της Κομισιόν ο οποίος δεύτερος κανονισμός ήρθε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης την οποία αμφισβήτησε ο πρώτος κανονισμός και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα γιατί να σας πιστέψουμε ότι έχετε τη βούληση να πάρετε επιτέλους μέτρα και να το χαριτολογήσω. Τι περιμένετε να σας κατατάξει, να κατατάξει την Κομισιόν κάποιος οίκος αξιολόγησης BB δεν ξέρω που θα σας πάει για να δράσετε να δείτε τον καταστροφικό ρόλο. Δεύτερο, για τα τεστ των τραπεζών. Γενικά περνάνε οι τράπεζες από εκεί. Με επιτυχία λένε. Μπορείτε να μου πείτε γιατί δεν ησυχάζουν οι αγορές και έχουμε κρίση χρέους. Μήπως οι αγορές θεωρούν ότι τα σενάρια κινδύνου που είναι στην ημερήσια διάταξη των τεστ είναι light. Δηλαδή να σας το πω πιο απλά, στα τεστ των τραπεζών μπαίνουν πιθανότητες, σενάρια, αυτά που κουβεντιάζουμε καθημερινά, κουβεντιάζονται, γράφονται στον τύπο, χρεοκοπίας της Ελλάδας, χρεοκοπίας της Πορτογαλίας, εξόδου από το ευρώ, τίθενται τέτοια σενάρια συζητιούνται αυτά στα, τεστ των τραπεζών. Και μια τελευταία για να μην σας κουράζω. Η ερώτηση τι θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρωζώνη δεν μου έχει απαντηθεί. Τι θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρωζώνη. Σας ρωτώ όμως ως Επίτροπος Ανταγωνισμού. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετέχει σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και ζητάει κάποια πράγματα. Ή κάνει τον κακό διαρθρωτικές αλλαγέ. Η ερώτηση είναι απλή. Πιστεύετε ότι οι απαιτήσει του διεθνού Νομισματικού Ταμείου στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μέσα στην κοινή αγορά. Αν έχετε κάνει τέτοια μελέτη θα με βοηθούσε πολύ να καταλάβω περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι και πάλι καλε διακοπέ. Okay, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν για τον κύριο Χοκμάρκ. Θα θέλω να επανέλθω στο να εξηγήσω ποιο είναι το μέσο που σκοπεύω να χρησιμοποιήσω για τις αποφάσεις αυτές του Δεκεμβρίου του Γενάρη. Δεν μιλάω για τη γενική στρατηγική όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό είναι πολύ ευρύτερο θέμα για τον Επίτροπο Ανταγωνισμού. Εγώ μιλάω για κάποια συγκεκριμένα θέματα, για τις αντιφάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Λόγω των σκέψεων για την αποτελεσματικότητα που συζητήσαμε προηγουμένως με κάποιους συναδέλφους, προσπαθούμε να βελτιώσουμε και κάποιες πτυχές της λειτουργίας των οικονομικών αυτών παραγόνων που προσφέρουν αυτές τις ε, γενικές υπηρεσίες στην αγορά, στις οικονομίες μας. Αυτό όμω είναι ένα τμήμα μόνο. Η ευρύτερη προσέγγιση, δούμε αυτό που ζητάμε στην Ευρώπη, είναι ότι έχουμε εδώ στην Ευρώπη ένα κατάλογο τομιακών διακανονισμών. Τομεί στου οποίου η υπηρεσία αυτή γενικού οικονομικού συμβαίνοντο είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Για τι τηλεπικοινωνίε, για την ενέργεια, για τι μεταφορέ, όλοι αυτοί οι διακανονισμοί γειτονιακοί είστε και εσείς νομοθέτες. Αυτές οι σκέψεις θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν. Ο έλεγχος των κρατικών ισχύσεων είναι ένα μέσο το οποίο εγώ προσπαθώ να το, να το εφαρμόσω κατά καλύτερα. Αλλά βέβαια δεν λύνει τα προβλήματα της οικονομίας μας, ε, τα προβλήματα αυτών που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, ε, το θέμα του ανταγωνισμού μέσα στην εσωτερική αγορά, ε, πέρα από την εσωτερική αγορά. Αυτό είναι τεράστια προβλήματα που θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με διάφορα μέσα που έχουμε που έχουν σαν στόχο να χρησιμοποιηθεί κατά τον ιδανικότερο δυνατό τρόπο το δημόσιο χρήμα, το χρήμα του φορολογούμενου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό ήθελα να τονίσω. Και προς τον κύριο Χουντή. Θα σας τα πω στα ισπανικά όμως. Ελπίζω ότι ε, όταν είμαι στην παραλία θα είμαι πιο ήσυχος, δεν θα μου υποβάλλουν τέτοιες ερωτήσεις συνεχώς. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα έχω χρόνο για να πάω στην παραλία, άλλο αυτό. Τώρα, οι υπηρεσίε αξιολόγηση, οι οργανισμοί αξιολόγηση μάλλον. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε δύο διαφορετικούς κανονισμούς. Στην αρχή της κρίσης, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πρώτη που εκφράστηκε για τους οργανισμούς αυτούς αξιολόγησης. Μετά υπήρχε μια δεύτερη φάση, στην οποία ληφθήκαν υπόψη και άλλες πτυχές. Αλλά ακόμα κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν πρέπει ακόμα να διακανονίσουμε κάποιες πτυχές. Και γι' αυτό προετοιμάζουμε ένα κανονισμό και δεν θα είναι και ο τελευταίος αυτός. Θέλουμε να παρεύουμε διακανονίζοντας κάποιες πτυχές και να διαγράψουμε κάποια άλλα σημεία από άλλους κανονισμούς, σημεία που αφορούν αυτούς τους οργανισμούς αξιολόγησης. Και θα πρέπει επίσης να ενδυναμώσουμε την αξιοπιστία όσον αφορά την δυνατότητα λήψης πολιτικών αποφάσεων για να ανεμετωστεί μια κρίση που είναι οικονομική αλλά έχει και πολιτικές πτυχές και μπορεί και να παρουσιάσει πάρα πολύ σημαντικά πολιτικά προβλήματα ούτως ώστε οι μηχανισμοί και η βάση λήψης αποφάσεων να είναι αξιόπιστοι και βάσιμοι. Γιατί βέβαια η αξιοπιστία των οργανισμών αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα εάν επιτρέψουμε πολύ ευραία περιθώρια λιγμών στις, ε, οργανισμούς αυτούς, θα έχουμε και τεράστια προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά τις ε, ε, τράπεζες και τις αρχές εποπτείας των τραπεζών, θα πρέπει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αυτές οι υπηρεσίες να συνεργαστούν όσον αφορά τα stress test θα δούμε τα αποτελέσματα την επόμενη Παρασκευή της 6 το απόγευμα. Πρέπει βέβαια να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και θα πρέπει να μπορούν οι αγορές να αντιμετωπίσουν την ευρικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ευθέας νομισματικό ταμείο. Υπάρχουν κοινά προγράμματα χρηματοδότησης και υποστήριξης. Και αυτά τα προγράμματα ισχύουν για τρεις χώρες στην Ευρώπη. Κοινή συνεργασία, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα πρέπει όμως να δούμε και ποιες θα είναι οι μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εισαγάγουμε. Και όσον αφορά παραδείγματος χάρη τις εθνικές υπηρεσίες ανταγωνισμού. Και χαίρομαι γιατί οι συνεργάτες μου συμμετείχαν στη συζήτηση των προγραμμάτων αυτών. και προσπάθησαν να συντονιστούν μεταξύ τους. Ε, τα προγράμματα αυτά είναι δύσκολα βέβαια να εφαρμοστούν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καλούνται και τα επιμέρους κράτη-μέλη να ενδυναμώσουν τις υπηρεσίες αυτές του ανταγωνισμού που έχουν και υπάρχουν και διατάξεις που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Αυτά από δική μου σκοπιάς, από σκοπιάς ανταγωνισμού δηλαδή, πρόεδρος. Τέλει και οι δύο υποβάλλοντας ερωτήσεις, Σόφιο Κόνη και Σίλβι Κούλακ. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ που έχετε έρθει εδώ στην Επιτροπή μας. Εγώ θα ήθελα να υποβάλω μια κάπως πιο γενική ερώτηση. Σε ορισμένους ε, τομείς, οι μόνοι, οι κύριοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ελόγου τομείς είναι οι κανόνες ανταγωνισμού. Παραδείγματος χάρη, αθλητισμός. Δεν υπάρχουν διατάξεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας που εφαρμόζονται συγκεκριμένα στον αθλητισμό. Απ' την άλλη μεριά, οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς, ιδίως οι κανόνες του ανταγωνισμού, εφαρμόζονται και στον αθλητικό κόσμο. Ε, όταν πρόκειται βέβαια για μια οικονομική δραστηριότητα προφανώς. Γι' αυτό η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωση σε αυτό τον τομέα, αλλά αυτό ισχύει και για άλλους τομεί και ιδιαίτερα για τι υπηρεσίε γενικού ενδιαφέροντο. Αυτή η πολιτική, λέω, διέπεται μόνο από τους κανόνες ανταγωνισμού, οι οποίε ε, δεν είναι πάντα διαφοροποιημένες τομέα παρόλο που ε, δικαστής μπορεί να, τις, να τους εφαρμόσει προσαρμόζοντας στον τομέα. Εγώ δεν έχω κάποιο... δεν παίρνω το μέρος κανένας εδώ στο θέα αυτό, αλλά θεωρούνται εσείς ικανοποιητικό, πολιτικά και νομικά, ότι οι ικανότητες ανταγωνισμού σε ορισμένου τομεί δεν αναφέρονται πάνω σε θετικές νομοθετικές διατάξεις που ορίζουν την αρμοδιότητα και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να επανέλθω στο παράδειγμα του αθλητισμού, πώς ορίζονται οι ε, ευρωπαϊκοί κανόνες ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στον αθλητισμό, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα ή σαφή πολιτική στον τομέα αυτών του αθλητισμού. Μπορείτε να μιλήσετε και στα Ισπανικά αν θέλετε στην απάντηση για να κάνω εξάσκηση στα Ισπανικά μου. Κύριε Πέτρο, σας ευχαριστώ που έχετε έρθει πολύ σύντομα, γιατί το, πρώτο, το κύριο ερώτημα που ήθελα να υποβάλω το υπέβαλε η Ελίζα Φερέρα, δεν θέλω να το επαναλάβω. Μια σύνομη λοιπόν παρατηρήση. Το Σώμα των Επιτροπών πρόσφατα αρνήθηκε να ε, νομοθετήσει όσον αφορά την πρόσβαση στι βασικέ τραπεζικέ υπηρεσίε και θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σα στο γεγονό ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ και ο κύριος Μπαντιά και ο κύριος Μπουζέκ αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό και πιστεύω ότι υπάρχει μια πτυχή ανταγωνισμού. Δηλαδή ε, εξασφαλίζουμε σε όλους τους ε, ενδεχόμενου χρήστε την πρόσβαση στι βασικέ τραπεζικέ υπηρεσίε, Αυτό είναι θέμα ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και θα μπορέσουμε να φροντίσουμε ούτω ώστε ε, τα τραπεζικά ιδρύματα να μην αρνούνται την πρόσβαση σε υπηρεσίες ε, το κάποιων πολιτών. Σας εύχομαι καλές διακοπές, αλλά θα έχουμε προβλήματα φαντάζομαι όλες στι διακοπές μας. Ευχαριστώ πολύ για το θέμα του αθλητισμού. Εάν καλά θυμάμαι στη νέα συνθήκη υπάρχει νέα νομική βάση. Δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί, αλλά υπάρχει νέα βάση για τον αθλητισμό. Από τη σκοπιά τη ανταγωνιστικότητα, του ανταγωνισμού μάλλον, υπήρξαν κάποιες σημαντικέ περιπτώσει, ιδίω για κάποια αθλήματα που έχουν επαγγελματική διάσταση και για τις οπτικοακουστικές τους προεκτάσεις υπήρξαν και οικονομικές, οικονομικά στοιχεία. Έτσι, ε, δεν είχαμε μεν τομεακέ κατευθυντήριε γραμμέ για κάποιες κρατικέ ενισχύσει, για την οικοδόμηση κρατικών υποδομών, αθλητικών, αλλά τις προάλλες μόλις συζητούσαμε υπεύθυνου υπηρεσιών μας για μια περίπτωση που μας απεσήμανε συγκεκριμένα η Ουγγαρία. Η Ουγγρική κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα χρηματοδότηση για την οικοδόμηση αθλητικών υποδομών, αθλητικών εγκαταστάσεων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ορισμένου επαγγελματικού ομίλου. Οπότε εκεί δημιουργείται θέμα επαγγελματικής, επαγγελματικού ανταγωνισμού. Είναι θέμα. Είναι πρόβλημα. Μα ζητούν με την κοινοποίησή του, μα ρωτούν μάλλον ε, υπό ποιε συνθήκε είναι συμβατή η βοήθεια αυτή με το πρόγραμμα κρατικών βοηθειών. Όπως για πολλούς άλλους τομείς ε, υπάρχουν κατευθυντήρες γραμμές μεν, αλλά για τις αθλητικές εγκαταστάσεις για πρώτη φορά δεν έχουμε απαραίτητο τι κατάλληλε κατευθυντήρε γραμμέ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την συνθήκη και να τη εφαρμόσουμε απευθεία ώστε να δούμε κατά πόσο είναι συμβατή, συμβατό το αίτημα της εγκουρικής κυβέρνησης με, ε, με το πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων. Και υπάρχουν και άλλες πτυχές του αθλητισμού που μπορεί να δημιουργήσουν θέματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό και ως προς την καταπολέμηση των ε, οικονομικών ομίλων, των τραστ. Ε, αν δεν κάνω λάθος όμως, η μόνη περίπτωση που συζητήσαμε ως σήμερα είχε να κάνει με τα οπτικοακουστικά δικαιώματα. Ήταν η οικονομική διάσταση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και σε άλλους τομείς υπάρχουν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκέ κατευθυντήρε γραμμές, δεν μα εμποδίζει να εφαρμόσουμε και του ευρωπαϊκού κανόνε και νόμου. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να ελέγξουμε τι κρατικέ ενισχύσει και για τα τράστια, και για τα καρτέλ και για τι συγχωνεύσει. Υπάρχουν σαφώ διαφορέ μεταξύ των χωρών κάποιες φορές κατά την υλοποίηση των κανόνων μας πρέπει να εξετάζουμε πώς εφαρμόζονται σε κάθε χώρα οι κανόνες. Ας σκεφτούμε τη Γαλλία. Η εξάλληψη του μονοπωλίου στο γαλλικό υπόδρομο, λόγω χάρη. Είναι μια ιδιαιτερότητα της Γαλλίας αυτή. Και έλεγα τις προάλλες τους συνεργάτες μου ότι είναι αδιανόητο πώς είναι οι Γάλλοι και οι Γαλλίδες που έρχονται να με δουν ή μου απέστειλαν επιστολές στη γειτονική. Σε μια γειτονική κιόλα χώρα, κανεί κανείς δεν μου απευθύνθηκε για το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα που αγγίζει τη Γαλλία. Εμάς φαίνεται πως όχι. Εγώ επιλήφθηκα του θέματος, αλλά πραγματικά υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες σε κάθε χώρα, διαφορετικοί τομείς με διαφορετικές ευαισθησίες. Κάποιες χώρες έχουν πολλές κατευθυντήρες γραμμές για κάποιους τομείς. Υπάρχουν πάνω από 30 γραμμές για διαφορετικούς τομείς και διαφορετικές κρατικές ενισχύσεις. Άλλε φορέ δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνε, οπότε εφαρμόζουμε απευθεία τη συνθήκη ή την ομολογία, όπω για τα τραστ, όπου έχουμε την απαραίτητη ομολογία. Εκεί καθορίζουμε την προσέγγιση μας ανάλογα με την περίπτωση τον τομέα. Πάντως, εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ασυμβατότητα. Δεν είναι ότι ο ανταγωνισμός ε, υπερκεράζει όλα τα υπόλοιπα. Όχι, χρειάζεται ο ανταγωνισμός, αλλά ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν αφήσουμε το κάθε κράτο να κάνει ό,τι θέλει, πάει η εσωτερική αγορά. Και τώρα για την ε, πρόσβαση στι βασικέ τραπεζικέ υπηρεσίε, κυρία Κουλέρ. Δεν είναι ότι υπάρχουν ε, φραγμοί για την ευρωπαϊκή νομοθεσία απαραίτητο. Από την άποψη του ανταγωνισμού, πρέπει να δούμε του φραγμού ω προ την αρχική πρόσβαση. Εκεί μπορεί να υπάρχουν θέματα ανταγωνισμού, αλλά δεν είμαι και βέβαιο ότι η πρόσβαση ενός ατόμου, ενός προσώπου σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να θεωρηθεί ως φραγμός που θα μπορούσε κανείς να τον ερμηνεύσει από την άποψη του ανταγωνισμού. Ε, κυρία ναι, αλλά σε σχέση με το τι μπορεί να συζητηθεί και στο κολέγιο Υπάρχουν τουλάχιστον 82 εκατομμύρια πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ένα πρόσωπο που έχει πρόβλημα πρόσβαση σε βασικέ τραπεζικέ υπηρεσίε, είναι εκατομμύρια. Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει και με τι επιχειρήσει που έχουν στην αγορά. Δεν είπα εγώ για τραστ. Ε, κοιτάξτε, ένα σύντομο ερώτημα έθεσα. Ε, άλλοι έχουν θέσει πέντε. Ε, ε, το σημειώνω, το σημειώνω και το καταγράφω. Ευχαριστούμε πραγματικά. Όπως είπα, θα σας ξαναδούμε στις 22 Σεπτεμβρίου. Όχι 22 Ιουλίου, όχι. Την γλιτώσατε. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και να συζητήσουμε τρεις τομείς της πολιτικής ανταγωνισμού. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας για αυτό το θέμα. Και υποτίθεται ότι θα έχει έρθει ο αντιπρόεδρο για να αναλάβει στη θέση μου. Οπότε θα πρέπει να ζητήσω στον επόμενο συνάδελφο, κατερχαιότητα, αρμόδιο, να αναλάβει. Όχι, είναι εδώ αντιπρόεδρο. Μισό λεπτάκι λοιπόν, μέχρι να έρθει ο συνάδελφο να αναλάβει την έδρα. Señorías, vamos a, continuar desarrollo normal de esta... Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Del que es ponente mi buen amigo και έλεγα ότι η εισηγητής είναι ο φίλος Ανδρέας Σφάμπ. Έχετε το λόγο κύριε Σφάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που σας άκουσα που μιλούσατε κύριε Πρόεδρε. Συζητούσαμε το θέμα της λογικής προσφυγής. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε αυτά τα θέματα σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα της λογικής προσφυγής ε, το συζητήσαμε και στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου και εγώ είχα την τιμή εκ μέρου τη Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων να ασχοληθώ με αυτή τη γνωμοδότηση μαζί με συναδέλφου ε, άλλων πολιτικών ομάδων. Τα είχαμε συζητήσει και στην οριζόντια ομάδα για το δίκαιο ανταγωνισμού. Το βασικό ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το αν ε, πρέπει να έχουμε ένα οριζόντιο εργαλείο και αν κάτι τέτοιο πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να καλύψει όλους τους νομοθετικούς ε, τομείς κατά εγκάρσιο τρόπο ή αν πρέπει να πούμε ότι επειδή αυτό το νομικό εργαλείο ε, μέχρι τώρα δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο, δηλαδή υπάρχουν ε, κάποιες χώρες που είναι περισσότερο προχωρημένες, αλλά γενικά δεν έχει εξελιχθεί πολύ αυτό το νομοθετικό εργαλείο στην ευρωπαϊκή νομολογία και μήπω γι' αυτό θα ήταν προτιμότερο να έχουμε ένα μικρότερο τομέα εφαρμογής σε μια πρώτη φάση που θα ασχοληθεί περισσότερο με τον, που θα εστιαστεί περισσότερο στον τομέα ανταγωνισμού είχε δώσει μια υπόσχεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και μέσω της πολιτικής ανταγωνισμού θα μπορούσαμε ε, να περάσουμε σε διαδικασία συναπόφασης ε, με βάση το άρθρο 114. Μέχρι τώρα ε, ε, είχαμε εξουσίες ε, τη Επιτροπής και του Συμβουλίου και μόνο γνωμοδοτήσεις του Κοινοβουλίου. Αν στον τομέα της συλλογική προσφυγή έχουμε θέματα πολιτική ανταγωνισμού, θα μπορούσαμε μέσω του άρθρου 114 να έχουμε διαδικασία συναπόφασης. Υπάρχουν βέβαια πολλά ανοιχτά θέματα και η πολιτική ομάδα του ΕΛΚ υπενθυμίζω ότι κάθε φορά τονίζει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην έχουμε αμερικάνικο κλίμα το οποίο θα επιβληθεί στην Ευρώπη. Είμαι πεπισμένος ότι ως Ευρωπαίοι νομοθέτες δεν έχουμε όλα τα απαραίτητα νομοθετικά εργαλεία για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργηθεί μια αμερικανική κατάσταση στην Ευρώπη. Και θα σας δώσω για παραδείγματα. Στην Γερμανία δεν υπάρχουν contingency fees, δηλαδή δεν συμμετέχουν ε, οι δικηγόροι στα ενδεχόμενα κέρδη μιας υπόθεσης. Παρ' όλα αυτά το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι στην περίπτωση που που ε, δεν έχει ο προσφεύγων μέσα για να ξεκινήσει μια προσφυγή θα μπορούσε σε περίπτωση επιτυχούς έκβαση της υπόθεσης ο δικηγόρος ε, να πληρώνεται από ε, τα ποσά που θα εκδικαστούν στην υπόθεση αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, σε ορισμένα κρατημέλη τουλάχιστον, θα μπορούσε να δημιουργήσει περιπτώσεις αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν στις ΗΠΑ με το σύστημα του class action, των συλλογικών προσφυγών στις ΗΠΑ. Και κατά αυτόν τον τρόπο ε, άμεσα μέσω του forum shopping, τη αναζήτησης δηλαδή του πιο βολικού δικαστηρίου, έχουμε μια διαφοροποίηση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο τομέι τη Νομολογία. και κατά τη γνώμη μου αυτό οδηγεί την δημιουργία ενός αμερικανικού συστήματος στην Ευρώπη, πράγμα το οποίο δεν θα επιθυμούσαμε. Όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη ε, είναι διστακτικά σε θέματα των συλλογικών προσφυγών και θα μπορούσαμε να, υποστηρίξουμε, να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν ε, στο εθνικό τους ε, αστικό δίκαιο τέτοιες ε, τροπολογίες που θα αφορούν τις συλλογικές προσφυγές και θα αποφεύγουν ένα αμερικανικό σύστημα συλλογικών προσφυγών. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν κάτι στο εθνικό του δίκαιο για να αποφύγουν το αμερικανικό σύστημα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα ήμασταν ανοιχτοί σε ένα σύστημα ε, ε, συλλογικών ε, προσφυγών για να μπορέσει να εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Ε, υπάρχουν συνάδελφοι, ο κ. Πρεσέντο και η κυρία Σόφι Ιντβέλ στην περασμένη θητεία του Κοινοβουλίου είχαν ασχοληθεί με αυτά και θα φέρω ένα παράδειγμα passing on defense ε, σε περιπτώσεις δηλαδή ε, που όταν αρχίζουν ε, περιπτώσεις ε, στρέβλωσης ανταγωνισμού μέχρι ε, τις τελικές επιπτώσεις τους καταναλωτές υπάρχουν πολλά στάδια και το ερώτημα θα ήταν αν μπορούμε μέσω αυτού του passing on defense να εφαρμόσουμε κάτι όσον αφορά ε, ε, τις απαιτήσει ε, από αυτόν ο οποίος ξεκίνησε την όλη διαδικασία. Υπάρχει επίσης το ερώτημα του πώς το ισχύον σύστημα της επικούς μεταχείρισης θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκάλυψη περισσότερων πληροφοριών προς την Επιτροπή είναι πληροφορίες που μπορεί να δώσει κάποιος και που σε μια κανονική υπόθεση ποτέ δεν θα έφταναν στη δημοσιότητα. Πρέπει να δούμε λοιπόν, ε, εξετάζοντας το σύστημα το οποίο ισχύει ε, και μόλι το ακούσαμε και από τον Επίτροπο Αλμούνια ότι μπορεί με το δίκαιο του ανταγωνισμού να καλύπτονται ορισμένε τέτοιε περιπτώσει. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω και ποια είναι η θέση των συναδέλφων από άλλε πολιτικές ομάδες ε, και σε λεπτομερή θέματα αλλά και ε, ω γενική προσέγγιση. Και μαζί με τι άλλε πολιτικέ ομάδε θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την γνωμοδότησή μα προ την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Τι θέλετε το ερώτημα και τη αρμόδια επιτροπή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Ο εισηγητής ε, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα και το παρουσίασε αναλυτικά. Όσον αφορά την ετήσια έκθεση υπάρχουν και οι νέες κρατικές ενισχύσεις και νέες προσεγγίσεις. Μπορείτε να αναφερθείτε και στις τρεις εκθέσεις. Ο κύριος Σίμων πρώτα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πάρω το λόγο για τη δική μου έκθεση πρωτοβουλίας, πρόεδρε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι αναφέρεται σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα η Κομισιόν. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη. Οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος ε, συμβάλλουν πάρα πολύ στο κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης, ε, στη ζωή των πολιτών και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Η προϋπόθεση για να λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες ιδανικά από σκοπιάς του πολίτη με υψηλή ποιότητα και ε, καθολική πρόσβαση για όλα τα στρώματα του πληθυσμού. Είναι πολύ σημαντικές προϋποθέσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες, πράγμα που προϋποθέτει ασφάλεια για εκείνους που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες και αυτούς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές όσον αφορά την νομική βάση, το νομικό πλαίσιο. Η πολύ καλή αξιολόγηση και διαβούλευση Κομισιών κατέδειξε όμως ότι εξακολουθεί να υπάρχει νομική ανασφάλεια και ανάγκη διευκρίνηση γιατί ακριβώς δεν υπάρχει το ζωστό ε, νομοθετικό πλαίσιο για τις υπηρεσίε αυτές. Το ανέφερε και προηγουμένω. θα πρέπει να εισαγάγουμε στη συζήτηση για λύση ενδεχόμενης ανασφάλειας ένα οριζόντιο νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες αυτές γενικού οικονομικού συμφέροντος βάσει του άρθρου 14. Με ένα τέτοιο οριζόντιο νομικό πλαίσιο δεν θέλουμε να παρέμβουμε στην προσφορά των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος αυτό η να είναι θέμα των κρατών μελών. Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο που θα δίνει τη δυνατότητα στις δημόσιες αρχές να ανταποκριθούν στις, ε, ε, στις ε, αρμοδιότητες τους, στις υποχρεώσεις τους μέσα σε αυτό το τομέα. Οι κανόνες ενισχύσεων είναι μόνο ένα τμήμα αυτού του ενδεχόμενου νομικού πλαισίου γιατί το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πολύ συγκεκριμένη νομοθεσία για κάποιες ε, νομοθετικές διατάξεις. Στην έκθεση πρωτοβουλίας που τελειοποιώ αύριο χαιρετίζουμε την ε, προσπάθεια της Κομισιόν να δημιουργήσει περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη βάση για την αξιολόγηση του θέματος των κρατικών ενισχύσεων στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Συγκεκριμένη προσέγγιση για να είναι τα πράγματα πιο απλά και να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια θα μπορούσαμε να φανταστούμε νύψωση των ε, κατοφλίων ή και εξαίρεση από την υποχρεώση κοινοποίησης. Ένας κανονισμός de minimis για υπηρεσίες πολύ περιορισμένης ε, τοπικής ε, εμβέλειας μου φαίνεται ότι θα ήταν κάτι καλό. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν επιπτώσει στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και εξασφαλίζεται έτσι ε, η μη ύπαρξη στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Όταν μελετήσουμε το θέμα νέων κανόνων de minimis για τις υπηρεσίες αυτές που είναι τοπικά περιορισμένες, θα μπορούσαμε να βρούμε μία προσέγγιση σε σχέση με το μέγεθος της ε, κοινότητας ή του Δήμου, τον αριθμό των ατόμων ή παραδείγματο χάνει των κύκλο εργασιών των λόγω επιχειρήσεων που προσφέρουν αυτή την ε, υπηρεσία. Συγκεκριμένα κατόφλια για κοινωνικές υπηρεσίες επίσης που δεν υπάρχει κίνδυνος στρέλπες στον νομισμού είναι μια δυνατή προσέγγιση εάν θέλουμε περισσότερη ε, διαφάνεια. Το ανέφερα και προηγουμένως. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν λογικό εδώ να συμπεριλάβουμε ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων ή ατόμων με ειδικέ ανάγκες να εξαιρεθούν από την υποχρεώση κοινοποίησης. Εάν από, ένα, ε, από έναν έλεγχο αποδειχθεί ότι υπάρχει συγκρισιμότητα με νοσοκομεία. Τέλος η Κομισιόν όσον αφορά τις μεγάλες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος βασίζεται στο ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες αυτές να προσφέρονται αποτελεσματικά. Είναι βάσιμο αυτό. Ε, διάβασα την περασμένη εβδομάδα όσον αφορά τις ενισχύσεις για τους γερμανικούς συνδρόμους για τη διατήρηση κάποιων σταθμών. Χωρίς έλεγχο, μόνο τους το χορηγούν, μόνο τους το ελέγχουν Γι' αυτό τίθεται το θέμα της νομικής βάσης. Και εγώ δεν βλέπω να υπάρχει μια νομική βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. στο άρθρο 106 θα ήταν η μόνη δυνατή νομική βάση. Τώρα έχουμε όμως την απόφαση Altmark του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και λέγεται εκεί ξεκάθαρα ότι αν υπάρχουν τέσσερα κριτήρια Altmark δεν υπάρχει καμία κρατική ενίσχυση. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή που θα μπορούσε να ελέγχει η Κομισιόν εφόσον πληρούν τα τέσσερα αυτά κριτήρια. Δεν προχωρήσαμε και πολύ στη συζήτηση προηγουμένως να αφορά το θέμα αυτό και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να βαθυνθεί στη συζήτηση των επόμενων εβδομάδων. <clears throat> θα πρέπει να ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή. Εγώ πάντως δεν βλέπω να υπάρχει νομική βάση για δράση της Κομισιόν σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σίμων. Ο Ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχουμε μια συζήτηση για τρία θέματα που έχουν σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού και ήδη κατά την συζήτηση με τον Επίτροπο εξέφρασα το ενδιαφέρον μου για τη συζήτηση στο, για το συγκεκριμένο θέμα των υπηρεσιών γενικών οικονομικού συμφέροντος. Εξέφρασα λοιπόν την ανησυχία μου για ένα θέμα που έχει να κάνει όχι μόνο με την επικουρικότητα, ώστε να μην καλύπτονται μόνο τα ζητήματα που έχουν κοινοτική διάσταση, αλλά και ένα σημείο που θα έπρεπε νομίζω οποιοδήποτε σχετικό νομοθέτημα να το καλύπτει. Θα έπρεπε εδώ να ευνοείται δηλαδή η συμπερίληψη της πρόσβασης στις υπηρεσίες και όχι να συμβαίνει το αντίθετο. Ε, να περάσω τώρα στην ε, στις συλλογικέ ε, προσφυγές που ανέφερε ο κύριος Σφάμπ και όπου θα πρέπει η δική μας Επιτροπή να υποβάλει σχετικά προτάσεις. Θεωρώ ότι είναι μείζονο σημασία στο θέμα αυτό για την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ιδίω σε ό,τι αφορά την διάσταση του ανταγωνισμού. Το έχουμε συζητήσει και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας και νομίζω ότι είχαμε καταλήξει σε κάποιες σημαντικές συμφωνίες όπως την αποτελεσματικότητα του κοινοτικού δικαίου, το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας που θεωρούσαμε καθοριστικό. Στον τομέα του ανταγωνισμού λοιπόν, λοιπόν υπάρχει νομολογία του δικαστηρίου που αφορά τις, ε, τα χρηματικά πρόστιμα και τις ποινές. Επίσης για τις ε, κατακατηγορία προσφυγές θα πρέπει και εδώ να λάβουμε υπόψη την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να δούμε κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία βεβαιότητας που θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη για την οικονομική διάσταση των περιπτώσεων. Να δούμε επίσης πώς μπορούμε να καλύψουμε και σε άλλους τομείς τις συλλογικές ε, προσφυγές. Πάντοτε ζητούσαμε να έχουμε κοινέ αρχές οριζόντιους κανόνες να αναζητούμε λύσεις συνεπείς που μόνο σε οριζόντιο επίπεδο μπορούν να εξευρεθούν από νομοθετικής βέβαια πλευράς. Φυσικά εδώ δεν υπάρχει πλήρη συμφωνία, αλλά νομίζω ότι ο γενικό προσανατολισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να οδεύσει προ την εναρμόνιση είναι καλή. Ένα λοιπόν νομοθετικό όργανο οριζόντιου χαρακτήρα σε αυτή τη χρονική φάση δεν θα ήταν τόσο λογικό, ακριβώ γιατί δεν υπάρχει και ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού. Για τι συλλογικέ λοιπόν συμβάσει, σε κάθε περίπτωση έχουμε να κάνουμε με εθνικέ διαδικασίε, με εθνικά δικαστικά συστήματα. Υπάρχουν διαφορετικές νομικές βάσεις και διαφορετικές αρμοδιότητες σε κάθε νομοθεσία. Υπάρχουν ε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Λόγου χάρη, τη στιγμή που κανείς υποβάλλει μια ε, προσφυγή συλλογική για κάποιο ελαττωματικό προϊόν, εδώ έχουμε τη σχέση του ε, ιδιώτη αγοραστή με τον πολιτή. Όμως, αν το δούμε από την άποψη του ανταγωνισμού, δεν μιλάμε μόνο για μια σχέση ιδιωτική, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε και με την με το ρόλο των δημοσίων αρχών στην ε, άσκηση των ευθυνών τους και στον, από τη σκοπιά του ανταγωνισμού. Δηλαδή, η άσκηση των αρμοδοτήτων των δημοσίων αρχών έρχονται πολλέ φορέ να επηρεάσουν και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί οι δύο τομείς είναι πολλέ φορέ αλληλένδετοι και συμπληρωματικοί. Εκεί λοιπόν απαιτείται η εξέβρεση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο τομέων, του ιδιωτικού και του δημόσιου. Έπειτα έχουμε και κάποια σχετική πείρα. Όλοι νομίζω συμμεριζόμαστε τα κριτήρια των ε, ακραίων φαινομένων του αμερικανικού προτύπου. Εάν συμφωνείτε εδώ, πολλές φορές μιλάμε για τριπλή αποζημίωση, ενώ εμείς το μόνο που θέλουμε είναι μια αποζημίωση που να καλύπτει την ε, υποβληθήσα ε, ζημία και να καλύπτει και τα προβλήματα που προκάλεσε μια ενδεχόμενη καθυστέρηση. Το τι συμβαίνει επίσης με τους δικηγόρους. Ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες η προσέγγιση είναι περισσότερο επικεντρωμένη στην ε, αλληλεγγύη. Εδώ θα πρέπει από την πλευρά του ανταγωνισμού σε, ευρωπαϊκή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διαφυλάξουμε και το στοιχείο εκείνο της επιγικίας που προβλέπετε και γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν μπορεί να παρέμβει κατά τρόπο δρασικό σε εθνικά συστήματα. Μιλάμε για συγκεκριμένα λοιπόν ζητήματα που θα πρέπει να τα δει κανεί ανά περίπτωση. Επίσης το πώς εξετάζονται οι προσφυγέ κατά κατηγορία στο αμερικανικό σύστημα. Εκεί πολλές φορές υπάρχουν και υπέρμετρες αντιδράσεις ή συνέπειες. Εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το δικό μας το σύστημα. Να μην υπονομεύσουμε την νομιμότητα των συλλογικών προσφυγών. Να υπάρχει λόγω χάρη συγκεκριμένη εντολή. Να μπορούμε να αναλάβουμε δράση υπέρ των θυμάτων, προς όφελος των θυμάτων. Αυτό ακριβώς ε, μας ενδιαφέρει κιόλα όταν υπάρχουν πολλά ε, θύματα ή ζημιοθέντες από μια συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν είναι και σημαντικό το πρόστιμο που θα επιβληθεί ακριβώ επειδή συγκεντρώθηκαν πολλοί μαζί προσφεύγοντε, τότε θα αποτραπούν και οι συμπεριφορέ που προκαλούν ακριβώ ε, τι ε, συμπεριφορέ τι αρχικέ. Και μα ενδιαφέρει και η προστασία των επιμέρους θυμάτων. Θα μπορούσαν λοιπόν να υπάρχουν ευρωπαϊκοί φορείς που να εξασφαλίζουν την εφαρμογή αυτού του συστήματος. Και εδώ χρειάζονται και εργαλεία διατομεακά, ώστε να υπάρχει και μια συνέπεια στο σύστημα συλλογικών προσφυγών. βλέπουμε ότι ακόμη και με την νομική μας βάση διαφέρει η θεσμική ισορροπία των σχέσεων που δημιουργούνται. Χρειάζεται λοιπόν κάποιες φορές μια ad hoc αποτίμηση του ε, βάρους που μπορεί να έχουν οι αποφάσεις μας από την πλευρά του ανταγωνισμού, ώστε να μην επηρεαστούν άλλοι τομείς. Θα πρέπει επίση να δούμε τι πείρα, τι γνώσει και τι πληροφορίε μπορούμε να αντλήσουμε από άλλου τομεί όπου υπάρχει ε, ένα πλούσιο πεδίο όπω σε αυτόν τον τομέα. Αλλά υπάρχουν άλλοι τομείς όπου σαφώς δεν υπάρχουν απαραίτητα ερευνητικά στοιχεία. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Ναι. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ήρθα εδώ όχι επειδή είμαι πιο σημαντικός από άλλους βουλευτές, αλλά επειδή είμαι ο πρεσβύτερος από τους η κυρία Οκονή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητέ Πίτερ, αγαπητέ συνάδελφε, καταρχήν χαίρομαι που η Κομισιόν ανέλαβε την ε, πρωτοβουλία να αναθεωρήσει τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Ξέρω ότι αυτό ήταν ένα αίτημα που είχε ε, υποβάλει η Επιτροπή ΕΚΟΝ όταν εξέτασε το θέμα της ε, γνωμοδότησης που από κοινού προετοιμάσαμε, Πέτερ, ακριβώς για τις ε, κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Εγώ συμμερίζομαι τις ε, πρωτοβουλίες που παρουσίασε ο Επίτροπος Αλμούνια για τη μεταρρύθμιση αυτή. Διευκρίνηση, πολύ σημαντικό στοιχείο, και διαφοροποιημένη και αναλογική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, πώς μπορούν αυτές οι δύο προτεραιότητες να ανεκατοπτριστούν σε ένα κείμενο. Συμφωνώ σε γενικές αμέσως με αυτά που είπε ο Πέτερ, αλλά έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Στο θέμα αυτό οι συζητήσεις είναι αρκετά συγκεχημένες συχνά. Ορισμένοι επιμένουν στην επικουρικότητα και θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αφήσει τις τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αρχές να ορίσουν τους κανόνες για τις δικές τους δημόσιες υπηρεσίες. Ορισμένοι βασίζουν την ιδέα αυτή της ε, επικουρικότητας σε μια πολύ πιο γενναιόδορη εικόνα των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος που θα πρέπει λένε να είναι ισότιμες με άλλες υπηρεσίες. Άλλοι του αντίον θεωρούν ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να ορίσουν ειδικού κανόνες, ξεφεύγοντας έτσι από τον κλασικό έλεγχο του ανταγωνισμού. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι πραγματική. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν πρέπει να φοβούμαστε την ευρωπαϊκή παρέμβαση. Του αντίον, ας είμαστε φιλόδοξοι ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να έχει μια νομική και πολιτική προσέγγιση συνεπή όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Αυτή η νομική προσέγγιση οπωσδήποτε περνάει, όχι μόνο όμως, από ένα καθεστώς ελέγχου των ε, κρατικών ενισχύσεων και θα ήθελα αυτή η μεταρρύθμιση να διευκρινίσει όλες τις ιδέες που παραμένουν ασαφείς είναι οικονομική δραστηριότητα ή όχι. Αυτό που είπες και εσύ Πέτερ. Α, ποιος, το, ποιος είναι ο φορέας, το περιφερειακό όφελος θα πρέπει για να μπορέσει να κρίνει κανένας να τοποθετηθεί στη θέση ενός τοπικού εκλεγμένου, κάποιου δηλαδή που γνωρίζει τους κανόνες και πρέπει να τους εφαρμόσει. Γι' αυτό πρότεινα την διατύπωση μιας μεθοδολογίας σαφούς, ακριβώς, που θα απευθύνεται προς τις ε, τοπικές αρχές και τις οργανωτικές αρχές, γιατί αυτή θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος ε, της μεταρρύθμισης. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε θα πρέπει να είναι χρήσιμο και πρακτικά εφαρμόσιμο για τις τοπικές αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Οκονή. Η Σοφίν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως πολλοί συζήτηση ε, πολλοί συνάδελφοι συγγνώμη παρακολουθώ τη συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε τις ίδιες συζητήσεις κάθε χρόνο τέτοια επιχειρήματα ίδιοι που παίρνουν το λόγο και εγώ μεταξύ αυτών και πάντα πριν από τις διακοπές τις ίδιες ανησυχίες εκφράζουμε συχνά όταν λέμε επικουρικότητα έχουν εντύπωση ότι δεν έχει καμία σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών αλλά έχει τα πάντα να κάνει με την ισχύ των πολιτικών. Θέλω να απομακρυνθούμε από αυτά και θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που η κυρία Κονού και ιδίω ο κύριο Σόκμαρ που δυστυχώ έφυγε. Δηλαδή θα πρέπει να αρχίσουμε τη συζήτηση για την ποιότητα και το μέλλον αυτών των υπηρεσιών. Βρίσκεται η Ευρώπη σε μια βαθιά κρίση. Είναι σαν να έχουμε παραλύσει, σαν να έχουμε αποσιωθεί και να βασιζόμαστε σε συστήματα του περασμένου αιώνα όχι συμπερινά. Πώς μπορούμε να κρατήσουμε τις ε, υπηρεσίες αυτές τα επίπεδα που έχουν σήμερα όταν δούμε ποιες είναι οι δαπάνες. Η δημόσια υγεία ξεπερνάει κάθε όρια. Δεν μπορούμε να πούμε θα κρατήσουμε τα πράγματα όσα έχουν. Δεν μπορούμε να μείνουμε στάσιμοι. Ο κόσμος ακολουθεί να γυρνά. Θα ήθελα λοιπόν, όπως είπε και ο Χόκμαρτ, να πάρω μια πιο οραματική, πιο τολμηρή στάση για όλα αυτά. Και κάποιες λεπτομέρειες που έθιξε ο εισηγητής κ. Σίμων όσον αφορά τα τεστ αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Δεν ξέρω κατά πόσο η έχει ή δεν έχει νομική βάση για να εξάσει την αποτελεσματικότητα. Εμένα δεν με νοιάζει. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι χρήστε των υπηρεσιών. Τι σκέφτονται. Γιατί οι υπηρεσίες δεν είναι για τη γραφειοκρατία, είναι για τους χρήστες. Θυμόσαστε όταν ήμουν εισηγήτρια για τη δέσμη, το... Θυμάστε τι είπε, θυμάστε, εντάξει, εντάξει, εντάξει, δεν είναι αστείο νομίζω. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό τι σκέφτεται η πολιτική για τις υπηρεσίες, είναι σημαντικό τι λένε οι χρήστες. Όταν εγώ το είχα προτείνω για δέσμη αντικρουστότε, ε, ε, θεωρήθηκε σαν ένα ανέκδοτο. Γιατί θεωρούσαν δηλαδή ότι αυτό που πιστεύουν οι χρήστες δεν είναι σημαντικό. Εγώ εξακολουθώ να έχω προβλήματα. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις αυτές, αναφερθήκατε στην ε, φροντίδα ηλικιωμένων παιδιών, ε, άτομα ειδικές ανάγκες, κοινωνική κατοικία κλπ. Βέβαια, ο στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι κοινωνικός. Το ίδιο ισχύει όμως και για τις δημόσιες μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες. Εγώ θα έλεγα ότι η πρόσφαση στη, στο διαδίκτυο ή στις τραπεζικές υπηρεσίες όπως έλεγχε προηγουμένως είναι σημαντικές για να μπορέσει κανένας να λειτουργεί τη σήμερα ως πολίτης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, προσφέρουν από τις δημόσιες αρχές. Άρα το ένα άλλο το άλλο. Και επαναλαμβάνω, όταν δω τις δαπάνες στον τομέα της δημόσιας υγείας, δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο όπως ε, τα περασμένα 50 χρόνια. Και οι κοινωνικέ κατοικίε στη χώρα μου είναι απελευθερωμένες. Υπάρχουν επίσης εκεί και εμπορικοί ε, ε, παράγοντες που προσφέρουν αυτή την, την υπηρεσία. Γιατί θα πρέπει αυτοί που είναι εμπορική. Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξαιρούνται από του κανόνες στον κόσμο. Σε άλλε χώρε είναι διαφορετικά τα πράγματα. δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε όλο το τομέα χωρί να εξετάσουμε εκάστοτε την πραγματικότητα. Δύο τελικά σχόλια. Πάντα όταν εξετάζουμε το θέμα της προσφοράς υπηρεσιών θα πρέπει να δούμε πάλι ποιο προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουν από δημόσια αρχή για να είναι καλέ. Οι δημόσιε αρχέ θα πρέπει να εξασφαλίσουν την προσφορά των υπηρεσιών. Συχνά δεν το κάνουν. Και τέλος, είτε προσφέρουν από δημόσιο ιδιωτικό παράγοντα ή κατά διαφορετικό τρόπο αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτό νομίζω και ο Χόκμαρ νομίζω είναι Ποια είναι τα κίνητρα κάποιου συγκεκριμένου τομέα για να βελτιωθεί η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και να μειωθεί και το κόστος. Αυτό είναι αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε. Και όχι κατά πόσο ο τομέα θα πρέπει να περιφερωθεί, να είναι δημόσιο ο προσφέρον την υπηρεσία ή όχι. Όχι. Θα πρέπει να έχουμε πάντα το φέρον των Χριστών κατά νου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Φιλίπ Λαμπέρτ έχει το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σοφή, δεν θα τσακωθούμε για μια φορά. Τίνω να συμβαδίζω με τη Σοφή και να λέω ότι δεν είναι άσπρο μαύρο και να πούμε είτε είναι κακή η αγορά και το κράτος είναι καλό ή το αντίστροφο. Και συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την οπτική γωνία του τελικού χρήστη. Αλλά ας ασχοληθούμε με τον τομέα της υγείας που ανέφερε. Στις ΗΠΑ Πολιτείες ε, το κόστος για την υγεία είναι 16% του ΑΕΠ και είναι ε, ε, κυρίως ιδιωτικοποιημένος ο τομέας. Στην Ευρώπη είναι 11% του ΑΕΠ το κόστος για την υγειονομική περίθαλψη και κυρίως είναι δημόσια υπηρεσία. Προσπαθώ λοιπόν ε, να κινηθώ προς την αποδοτικότητα και να δω ποιο είναι, ε, το όφελος που έχω για τα χρήματά μου και ε, το αποτέλεσμα με μετρήσιμα αποτελέσματα προσδόκιμο επιβίωσης, ποιότητα ζωής κλπ. δείχνουν ότι εμείς με 11% του ΑΕΠ στην Ευρώπη κυρίως στα, χέρια του δημοσίου, πάμε καλύτερα από ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε με μεγαλύτερη δαπάνη. Γι' αυτό επιλέγω εγώ ένα δημόσιο σύστημα έναντι ενό ιδιωτικού. Υπάρχει εδώ σπατάλη πόρων Προφανώς και υπάρχει σπατάλη πόρων και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την απόδοση του συστήματος και εδώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά γνωρίζω αρκετά καλά τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορώ να πω ότι υπάρχουν και στον ιδιωτικό τομέα σπατάλε και εκεί υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικότητα. Και αυτό το οποίο με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι όταν εξετάζει του περισσότερου ιδιωτικού φορεί, γιατί αν έχει ασχοληθεί με το θέμα το ξέρει, ο τελικό χρήστη, ο πελάτη, ε, έρχεται υπαριθμό 3 ή υπαριθμό 4 ω ε, ε, ως μέλημα για τις εταιρείες. Το, στις πρώτες θέσεις είναι ο μέτοχος και μόνο ο μέτοχος. Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι εις βάρος του τελικού χρήστη. Ας μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν, ας μην νομίζουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας θέλει να βελτιστοποιήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ε, με το ελάχιστο κόστος. Ο στόχος του ιδιωτικού τομέα που κοντόφθαλμα το εξετάζει είναι ότι θέλει να εξασφαλίσει κέρδη για τους μετόχους. Δεν λέω ότι είναι λάθος το να έχουν κέρδη για τους μετόχους, αλλά αν αυτή είναι η βασική προτεραιότητα, τα κέρδη των μετόχων, έτσι έχουν τα πράγματα. Ακούω πολλούς που λένε ότι δεν έχει καλή απόδοση ο δημόσιος τομέας. Αυτό όμως που θέλουμε εμεί δεν είναι να λάβουμε υπόψη μας κατά κύριο λόγο τους μετόχους των, μεγάλων, των πολύ μεγάλων εταιριών, γιατί όλο προ εκεί κινούμεθα. Εγώ γνωρίζω τη χώρα μου και ξέρω ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση σχετικά ε, με τα κέρδη των ιδιωτικών εταιριών. Ε, αλλά δεν ε, θέλω να είναι ο στόχος μας η μεγιστοποίηση του κέρδους για τους ε, μετόχους τους οποίους δεν μπορούμε να έχουμε ε, ρυθμιστική πρόσβαση. πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα της νομικής βάσης ε, που ανέφερες, αλλά νομίζω ότι αυτό που μας χρειάζεται είναι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τις ε, υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και αυτό το οποίο κάνει ο κ. Σαλμούνια και η Γενική Διεύθυνση Επιτροπής νομίζω ότι είναι θετική και προς τον Πέτερ Σίμων θέλω να πω ότι μου αρέσει η προσέγγιση σας και πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε απλούς κανόνες θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αν δεν υπάρχει στρέβλωση της αγοράς ή αν εξετάζουμε κάποιο μικρό επίπεδο όπως το επίπεδο της τοπικής περιφερειακής αγοράς που δεν επιφέρει στρέβλωση στην αγορά ε, να δίνουμε πιο εύκολα την έγκρισή μας. δεν λέω να έχουμε ε, ένα γενικό σύστημα για όλους, αλλά όσο δυνατόν απλούστερο, γιατί αν το κάνουμε πιο σύνθετο το σύστημα, δημιουργούνται περισσότερες παρανοήσεις. Ε, Ανδρέας, ξέρω ότι ε, συμφωνείς και εσύ με τις ανησυχίες που έχω όσον αφορά την ε, έκθεση για τον ανταγωνισμό μερικές φορές νομίζω ότι κάνουμε τα πράγματα κατά συνήθεια χωρίς να προσπαθήσουμε να αποκομίσουμε κάποιο όφελο, Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε. Να πούμε ότι αφού δεν ακούγεται η γνώμη μας να μην ξανακάνουμε έκθεση ή να κάνουμε μια έκθεση με ένα άρθρο και μόνο και να πούμε ότι αφού δεν μας ακούτε δεν χρειάζεται να ξαναπούμε κι εμείς τίποτα γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε αποδοτικότητα της ενέργειας και θα διαφυλάξουμε την ενέργειά μας για κάτι σημαντικότερο και αποδοτικότερο. Προτείνω μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια πιο έξυπνη ιδέα για να μην μείνουμε στα ίδια και τα ίδια γιατί ε, θα ξαναλέμε τα ίδια πράγματα που θα παραμένουν νεκρό γράμμα, πράγμα το οποίο δεν ε, επιθυμούμε και αφήνω τα θέματα συλλογικής προσφυγής στους άλλους συναδέλφους. Ευχαριστούμε, Φιλίπ, Πρόεδρος. Σε απάντηση σε αυτά που είπες, Φιλίπ, νομίζω ότι ε, για την έκθεση αυτή είπαμε ότι θα κάνουμε μια έκθεση γιατί ε, θέλουμε όχι απλώς να αντιδρούμε στην έκθεση της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό, αλλά να υποβάλουμε τη δική μας έκθεση για τον ανταγωνισμό με αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε σκόπιμο να πούμε για τον, πούμε για τον ανταγωνισμό. Σόφη, ήθελε το λόγο, αλλά έχω ακόμη άλλου τέσσερι ομιλητέ και βέβαια και πρέπει οι δύο εισηγητέ να λάβουν το λόγο. Αλλά ξέρω ότι από αυτά που είπε ο Φιλίπ, κάτι σου κίνησε την προσοχή και θέλει να απαντήσει. Ε, να διορθώσω μια παρανόηση, λέει η κυρία Ινβέλτ. Δεν είπα ότι πρέπει ή δεν πρέπει να, να απελευθερωθεί κάποιο τομέα. Είπα ότι πρέπει να εξετάσουμε τα κίνητρα σε συγκεκριμένου τομεί για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και το κόστο. Η συζήτηση αυτή συνεχώς στρέφεται γύρω από το αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κρατικές ενισχύσεις οι δημόσιες αρχές. Και εγώ θέλω να βάλουμε το θέμα της αποδοτικότητας και του κόστους μέσα στη συζήτηση. Δεν μιλώ για απελευθέρωση του τομέα ή όχι. Ωραία. Ο Σφεν, ο κύριος Κυλακάκης και μετά πάλι ο Πέντε Σίμων και ο Ανδρέας Σφάμπ. Ο Σβέν. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα είμαι σύντομος για το θέμα των συλλογικών προσφυγών ή το θέμα ε, των ε, συμπράξεων στον τομέα των προσφυγών όπως ε, με φρικτό τρόπο το αναφέρουν οι νομικοί. Το θέμα είναι αν είναι θέμα της Οικονομικής Επιτροπής. Δηλαδή έχουμε εδώ τομείς στους οποίους πολλοί πολίτες μπορεί να έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, προβλήματα και με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ε, και θέλουμε να εκπροσωπούνται τα συμφέροντα των καταναλωτών σωστά και γι' αυτό θέλουμε να δυναμώσουμε εμείς συγκεκριμένους τομείς. Μπορεί σε συγκεκριμένε περιπτώσει, δηλαδή, κάποιο, ένα πολίτη από μόνο του, να μην μπορεί ε, να αντέξει το βάρο τη κίνηση τη διαδικασία προσφυγή αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλές δυνατότητες ε, ε, κατάχρησης ε, σε πολλά κράτη-μέλη είναι τόσο υψηλά τα, τα στοιχεία κόστους ασφάλειας που δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι για να κινηθεί σε ένα τομέα. Και ξέρουμε ότι πολλοί δεν θέλουν να ασχοληθούν καθόλου με το θέμα των συλλογικών προσφυγών Υπάρχουν πολλοί, πολλές ομάδες άσκησης ε, πίεσης και πολύ συχνά λέγεται ε, ας κάνουμε μια πρόταση που θα ισχύει για όλους τους τομείς, γιατί αυτό θα ήταν η καλύτερη μέθοδος για να βρούμε τη σωστή προσέγγιση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι προ όφελο των καταναλωτών, γιατί κάθε χρόνο οι καταναλωτέ θίγονται σε ύψο δισεκατομμυρίων. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα και δεν πρέπει να το αφήσουμε κατά μέρο. Και η εκπροσώπηση των καταναλωτών ε, από νομική πλευρά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενισχύσουμε και πρέπει να το εξετάσουμε και κατά οριζόντιο τρόπο. Παράλληλα, ίσω είναι σκόπιμο να κάνουμε προτάσεις που θα είναι συγκεκριμένε ανατομέα, ούτως ώστε να έχουμε κάποια δυνατότητα να κερδίσουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προσφυγών. Ο ρόλος των οργανώσεων καταναλωτών σε αυτό το τομέα πρέπει να ενισχυθεί και να περιορίσουμε τις περιπτώσεις καταχρήσεων και μπορούμε να βρούμε περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να ασκηθούν συλλογικές ε, προσφυγές, ε, συλλογικών προσφυγών, στις οποίες δεν τίθεται θέμα προστασίας του καταναλωτού, αλλά απλώς τίθεται θέμα ε, αποκόμισης του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους. Και αυτές τις δύο περιπτώσεις πρέπει να τις διαχωρίσουμε. εν ολίγης, ε, συμφωνώ να έχουμε μια οριζόντια ε, προσπάθεια για τις λογικές προσφυγές, αλλά τα μέτρα τα οποία θα προτείνουμε θα πρέπει να τα διατυπώσουμε με έξυπνο τρόπο, τρόπο ώστε να ε, επωφελούνται αυτοί που πρέπει να υποφεληθούν γιατί πολύ συχνά μπορεί να χάσουμε από το κατάλληλο πεδίο αυτούς που πραγματικά είναι υπεύθυνοι. η Επιτροπή μας είπε ότι μπορεί να μην έχουμε ε, μία περιοριστική ρύθμιση αλλά απλώς ε, μία σύσταση ε, σε διάφορους τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όπως διάφοροι τραπεζικοί λογαριασμοί και με την ενίσχυση των δυνατοτήτων για τις συλλογικές ε, ε, προσφυγές θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι υπέρ των καταναλωτών ε, στην Ευρώπη και όχι υπέρ των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων. μια εταιρεία έχει μεγάλο κεφάλαιο και σαφώς έχει πλεονέκτημα πληροφόρησης ε, έναντι των ε, πολιτών ε, και θα πρέπει να προσφέρουμε στους καταναλωτές αυτό το οποίο κατά περίπτωση χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κυλακάκης. Κυλακάκης. Thank you, yes. Madam President. I, I have a double problem here. I can't read it that. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπορώ ούτε να διαβάσω τόσο μακριά το ταμπελάκι και δεν διαβάζω και εδώ καθαρά αυτό που έχω μπροστά μου. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αναφορά στο αμερικανικό σύστημα υγείας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι το σύστημα υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών υποφέρει με την εσωτερική ζήτηση η οποία είναι μια ιδιαιτερότητα του συστήματος αυτού του υγειονομικού σε κάθε περίπτωση. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε ξεχωριστά και ως μια εξαίρεση σε όλες τις χώρες. Οι ανεπάρκειες των αγορών που συζητούμε πρέπει να παραλληλιστούν προς τις ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος. Και επειδή είμαι Έλληνα πρέπει να σας πω ότι οι ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρέ από τις ελλείψει των αγορών. Ιδίω αν αυτές τι ανεπάρκειες δεν τις αντιμετωπίσει κανείς ε, εγκαίρω. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια πιο εξελιγμένη προσέγγιση εδώ, γιατί τα πολιτικά συστήματα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης δεν λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορούμε να, δεν να θεωρούμε την προστασία των καταναλωτών ταυτόσιμη σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί να ισχύουν οι ίδιοι κανόνε όπου υπάρχει μια ισχυρή θεσμική προστασία ή προσέγγιση εντό του δεδομένου κράτου αλλά το συγκεκριμένο κράτος έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση προς όλους αυτούς τους τομείς λήψης αποφάσεων πολιτικών. Ξέρουμε ότι οι αγορές έχουν ανεπάρκειες παρόμοιες παντού, όμως τα πολιτικά συστήματα διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πολύ σύντομα για το θέμα των συλλογικών προσφυγών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προς υπάρχει μια πρόταση ότι εκείνοι που εργάζονται στο News of the World μπορούν να ζητήσουν συλλογική προσφυγή γιατί έχουν στιγματιστεί από, κάποιες, ε, από κάποια συμβάντα. Ε, δεν είναι πρώτο φανέ αυτό. Υπάρχουν προηγούμενα. Γιατί εκεί καμιά φορά έχουμε συλλογέ προσφυγέ εκεί που δεν τι περιμένουμε. Τώρα θέλω έρθω στου δύο συζητητέ, Πίτερ Σίμον και μετά Ανδρέα. Ja, also ich muss Sophie äh, recht geben. Έχει δίκιο η Σοφή. Κάθε χρόνο κάνουμε την ίδια συζήτηση. Με τα ίδια άτομα και τα ίδια επιχειρήματα. Και λυπάμαι που δεν θα πρόκειται να συναντηθούμε ποτέ στι απόψει ακόμη και αν είμαστε 20 χρόνια εδώ. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Εγώ δεν ήθελα να κάνω αυτή τη συζήτηση επί τη ουσία. Γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή και εδώ. Το μόνο που πρέπει να εξετάσουμε σήμερα είναι η μεταρρύθμιση των διατάξεων ε, κρατικών ενισχύσεων για το οποίο είναι αρμόδιος ο ανταγωνισμός και έχει ορίσει όρια το ΔΕΚ τι είναι και τι δεν είναι κρατική ενίσχυση και όταν συζητάμε το θέμα της απορρισματικότητας η βελτίωση της ε, ε, προσφοράς για τους πολίτες και όλα αυτά θέλουμε να το σε αυτό το πλαίσιο τότε θα πρέπει να πούμε στην Κομισιόν όπως το έκανα και προηγουμένως ότι εντάξει θα το συζητήσουμε εφόσον υπάρχει μια νομική βάση. Ε, όσο δεν υπάρχει όμως νομική βάση και ακριβώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφαση Άλμακ είπε πότε δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση, πότε δεν υπάρχει δηλαδή αρνητικότητα της Κομισιόν για να διακανονίσει. Εμείς ως κοινοβούλοι που πρέπει να ασκήσουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Κομισιόν δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τη θεματοφύλακα των ε, συνθήκων «Α, δεν μας νοιάζει αν έχετε αρμοδιότητα ή όχι, κάντε εκεί από αυτό που σας λέμε». Μα δεν γίνεται αυτό και γι' αυτό αναγκάστηκα να γελάσω εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν μας νοιάζει αν υπάρχει νομική βάση ή όχι. Γιατί εάν εδώ στο πρωτογενές ή δευτερογενές ε, δίκαιο έχουμε αρμοδιότητα, είναι ένα θέμα. Αν δεν έχουμε, ας τη δημιουργήσουμε τότε. We're getting so passionate the... Ευχαριστώ πολύ, αλλά Μιλάτε τόσο γρήγορα στον ενθουσιασμό σα που δεν σα προλαβαίνουν η διερμηνής. Ο κύριο Σβάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την έκθεση του συναδέλφου Σίμων, καταρχήν, όπως είπε και η Σοφία Οκονή, πιστεύω ότι έχει δίκιο, ε, πρέπει να κάνουμε κάτι και εμείς από πλευράς ε, του ΕΛΚ θα ε, ε, κάνουμε κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Και έχει δίκιο και η συνάδελφος Σοφή Ιντβέλντ σχετικά με την κατάσταση στην Ευρώπη και την αποτελεσματικότητα. Δεν αποκλίνουμε λοιπόν αυτό το θέμα της αποτελεσματικότητας, αλλά εδώ συμφωνώ με τον συνάδελφο Σίμων ότι πρέπει να βρούμε τη σωστή νομική βάση. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Το θέμα είναι αν αυτή η απόφαση ε, Altmark ε, ε, πρέπει να, πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα αυτών τα οποία κάνουμε και σε τι βαθμό μπορεί να ασκήσει τον έλεγχο η Επιτροπή. νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε μια οδηγία πλαίσιο με βάση άρθρο 14 σε σχέση με αυτό που είπε ο συνάδελφο Σίμων. Ε, ήταν ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του συναδέλφου Λάμπερτ σχετικά με την υποβολή εκθέσεων Μα ενδιαφέρει το πώ θα διαμορφώνονται οι εκθέσει αυτές στο μέλλον για να μπορέσουμε εποφελώ ε, να ασχοληθούμε με αυτές τις εκθέσει ε, για την ανταγωνιστικότητα και αυτό θα κάνουμε και κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Περνάω τώρα στο θέμα της, ε, των συλλογικών προσφυγών θέλουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους που αναφέρετε και πρέπει να δούμε με τι τρόπο θα, του, θα τους επιτύχουμε. Και η κοινή εκπροσώπηση είναι κάτι το οποίο είναι ε, απαραίτητο ενώ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και ο συνάδελφος Σάντσες Προσέντο μίλησε για την οικονομία της διαδικασίας. Νομίζω ότι και αυτό συνάδει με την κατεύθυνση ε, ε, ε, της του να επιτρέπουμε τις λογικές προσφυγές. Και στη Γερμανία αυτό έχει σχέση με την υπόθεση για την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. να δούμε ε, ε, ε, αυτό που αν κάτι μπορεί να εφαρμοστεί στο χρηματοπιστωτικό τομέα και κατά πόσο μπορούμε να το μεταφέρουμε και σε, και σε άλλους τομείς. Τίθεται το ερώτημα αν συμφωνούμε ότι πλήττονται τα συμφέροντα των καταναλωτών και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη δυνατότητα της λογικής προσφυγής το ερώτημα τίθεται ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής, γιατί η Επιτροπή, τον διακόπτει η Πρόεδρος στον ομιλητή, Ε, παρακαλώ να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει η Πρόεδρο. Πάντω, χρειαζόμαστε, κύριο Σφαμπ, ε, ένα σαφέ πλαίσιο ε, για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αυτεπαγγέλτο μπορεί κάτι να ρυθμίσει και από την άλλη μεριά ιδιωτικών προσφυγών που μπορούν να κατατεθούν. Πάντω, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Μια συζήτηση που νομίζω θα ενθουσιάσει όλου του ειδικού κατά του επόμενου μήνε. Έχουμε το χρόνο τώρα το καλοκαίρι για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και να ξεκουραστούμε έχοντα και αυτά που σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λένε ότι έχουν μια παρατήρηση για την νομική βάση. Παρακαλούμε πολύ σύντομα. Σε 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με την νομική βάση για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, Σύμφωνα με την απόφαση Altmark και ό, αν, αν όλα τα κριτήρια της απόφασης αυτής πληρούνται, αποζημίωση για αποτελεσματική επιχείρηση δεν είναι ενίσχυση. Ένα τεστ αποδοτικότητας δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, αλλά να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη, να λάβουν υπόψη την αποζημίωσή τους, την αποτελεσματικότητα, ώστε να ενθαρρύνουν τους φορείς της αγοράς να είναι πιο αποδοτικοί, πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστούμε. Εάν οι συγητέ χρειαστούν περισσότερη βοήθεια, θα σα ζητήσουν τι απαραίτητε πληροφορίε. Τώρα το χρονοδιάγραμμα για τι εκθέσει αυτέ. Η ετήσια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισμού, υποβολή τροπολογιών στι 30 Σεπτεμβρίου, εξέταση στις 17 Οκτωβρίου, ώστε να ψηφίσουμε στις 22 Νοεμβρίου. Και να περάσει στη δεύτερη ολομέλεια του Δεκεμβρίου το θέμα αυτό, η μεταρρύθμιση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, υποβολή τροπολογιών στις 15 Σεπτεμβρίου, εξέταση στις 3 Οκτωβρίου, 4 Οκτωβρίου ψηφοφορία και θα περάσει στην ολομέλεια, τη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου ελπίζουμε. Έπειτα η έκθεση για τη συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση στις συλλογικές προσφυγές ε, ακρόαση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στις 22 Σεπτεμβρίου, υποβολή τροπολογιών στις 23 Σεπτεμβρίου, εξέταση των τροπολογιών 4 Οκτωβρίου, ψηφοφορία την ίδια μέρα, 4 δηλαδή Οκτωβρίου, και στόχος μας να περάσει στην πρώτη Ολομέλεια του, Οκτω... Νοεμβρίου. Νομίζω αυτό ικανοποιεί τις ανάγκες του χρονοδιαγράμματος της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ και περνάμε τώρα στο σημείο 12 σχέδιο έκθεση τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού του 2012. Εισηγητή ο κ. Λούμπιξον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Μπαλτζάνη που είναι καθήλυν αρμόδια συγγήτρια για, το, για την έκθεση αυτή που παρουσιάζω σήμερα. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να τις καταστήσω σε αυτή τη δική μας θέση για τον προπολογισμό του 2012. Βρισκόμαστε στην τελευταία φάση της συζήτησης στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων για τον προπολογισμό αυτό εδώ έχουμε να κάνουμε με πολιτικούς προσανατολισμούς και με συγκεκριμένα ποσά. Κατά την άποψή μου πρέπει να διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες θεμάτων αυτά που μας απασχολούν. Πρώτα απ' όλα την πολιτική μας, την πολιτική μας τάση και έπειτα το έγγραφο εργασίας όπου θα επικεντρωθούμε στους αριθμούς. Στο έγγραφο εργασίας Έχουμε μια αναθεωρημένη εκδοχή που τη λάβαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χθες το βράδυ. Θα το βρείτε αυτό στο φακελό σας. Εγώ φρόντισα να, να ενημερώσω τα στοιχεία αυτά μετά την προκατακτική παρουσίαση από το Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχουν εκεί προτάσεις μείωσης σε πολλούς τομείς. Στο έγγραφο εργασίας ε, το επικυρωποιημένο φρόντισα να συμπεριληφθούν τροπολογίες σε σχέση με τους αριθμούς, τα ποσά που προτείνει το Συμβούλιο. Ωστόσο, για τις πολιτικές προτεραιότητες που αναφέρονται δεν επιφέραμε έλεγε. Εγώ επικεντρώθηκα σε τέσσερις τομείς. Συγκεκριμένα την καταπολέμηση της απάτης, της φοροδιαφυγής, την, ε, τον έλεγχο την ε, επίβλεψη και την ανάκαμψη, ώστε να ξαναβρούμε σταθερότητα οικονομική στην Ευρώπη. Είναι σαφές ότι οι ευρωπαϊκές ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να έχουν ε, απαραίτητα αναγκαία κονδύλια ώστε να γίνουν ανεξάρτητος φορέας και παράγοντας της αγοράς. Σε αυτή τη φάση της, αναδιάρθρωσης, της προσπάθειας αναδιάρθρωσης είναι δύσκολο κάτι τέτοιο θα πρέπει να στηριχθούν οι αρχές αυτές, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρξει και αύξηση των κονδυλίων. Εφόσον αυξάνονται οι ευθύνε τους, πρέπει να αυξηθούν και οι πόροι τους. Υπάρχει εδώ πρόταση του Συμβουλίου που οδεύει προς την αντίθετη κατεύθυνση, με περικοπές, με μειώσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να πούμε όχι, όχι σε αυτές τις προτάσεις. Πρέπει επίσης να υπάρξει βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης. Στο επίπεδο της Επιτροπής πρέπει να εξευρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να μπορεί κανείς να επιθεωρεί επαρκώς την δημοσιονομική και φορολογική κατάσταση των κρατών Χρειάζεται περισσότερο προσωπικό ε, σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΦΙΝ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αναδίπλωση του προσωπικού. Δεν είναι η λύση αυτή. Πώς θα τα καταφέρουμε όταν θα υπάρξουν τα νέα μέτρα από το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης που θα χρειαστούν υλοποίηση. Χρειάζεται προσωπικό με τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, ώστε να μπορεί να εξεύρει και λύσεις στα προβλήματα. Εδώ πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, που θα έχουμε στο προσεχές χρονικό διάστημα για τα στατιστικά δεδομένα. Εδώ δεν υπήρξαν επαρκείς προτεραιότητες. Ε, έχει γίνει σαφές ότι η ποιότητα, ε, η έκταση των δεδομένων πρέπει να βελτιωθεί ανά περίπτωση και για να είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα από την όλη προσπάθεια. Εάν οι θέσει του προπολογισμού που τώρα προβλέπονται, τα ποσά δηλαδή δεν επαρκούν, πρέπει να αυξηθούν. Το Συμβούλιο όμω οδεύει προ την αντίθετη κατεύθυνση πάλι. Προτείνει και εδώ μείωση, περικοπέ στον προπολογισμό για τι στατιστικέ. Κατά τέταρτο, η καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει έλεγχο εντελεχή. Η κρίση μα απέδειξε ότι Χρειαζόμαστε αποτελεσματικά συστήματα συλλογής των φόρων. Εδώ πρέπει να αυξηθούν οι πόροι και της Γενικής Διεύθυνσης ε, των Φορολογικών Θεμάτων. Δεν συμφωνώ καθόλου με την πρόθεση του Συμβουλίου να προχωρήσει σε μειώσεις, ούτε σε αυτό το τομέα. Ως σήμερα οι συζητήσεις ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικές ε, στην Επιτροπή μας Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Ελπίζω ότι έτσι θα προχωρήσουμε και ως την ψηφοφορία του φθινοπόρου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον Ζαν Πολ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω τα κύρια θέματα που έθιξε ο εισηγητή είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το παράδοξο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ότι τα κράτη-μέλη θέλουν ο ευρωπαϊκός προπολογισμό να είναι αυστηρός, λιτός, νόμιμο, αλλά να μην υποστεί τις επιπτώσεις των απαραίτητων επιπτω... από των τροποποιήσεων της χορήγησης των πορών από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δεν μπορεί να θέλουμε και περισσότερη υποπτία και πραγματική οικονομική διακυβέρνηση χωρίς να δώσουμε και τους απαραίτητους τα απαραίτητα μέσα. Λοιπόν, δεν μπορούμε στους τομείς αυτούς να μειώσουμε τους πόρους σημαντικά. Αν πάρω το ΕΣΜΑ, είμαστε στο Παρίσι χθε για να εγκατασταθεί στους, στους, νέα γραφεία και να αναλάβει τις ε, επίσημες ε, ε, ευθύνες του, αλλά πολλές καλές προθέσεις χωρίς επαρκή μέσα, ούτε οικονομικά, ούτε ανθρώπινα, ούτε τίποτα. Και θέλω να σας πω ότι όλοι μιλάνε για τις υπηρεσίες αξιολόγησης, οργανισμούς αξιολόγησης, σήμερα το πρωί είπαμε 20 φορές. Κανένας δεν τόνισε όμως ότι καμιά από τους ε, οργανισμούς αυτούς ε, αξιολόγησης, τις τρεις μεγάλες αυτές, δεν είναι εγκεκριμένε ούτε ελέγχονται. Υπάρχουν λόγω της ρήτρα του παππού, όπως λέγεται, επειδή υπήρχαν στο παρελθόν. Δηλαδή, οι αρχές που είναι υπεύθυνε για να συγκρίσουν δεν έχουν ούτε χρόνο ούτε τη δυνατότητα για να για να τις ελέγξουν. Τα κάνουν δηλαδή όπως για την κοινωνική ασφάλιση στη Γαλλία που όταν δεν έχει το κράτος να πληρώσει λέει «Α, λείπουν τα δικαιολογητικά σας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Γι' αυτό ακριβώς εγώ και το ΕΛΚ υποστηρίζουμε τις προτάσεις του εισηγητή που είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Ταυτόχρονα όσον αφορά τις στατιστικές, όταν δούμε σήμερα τη σημασία τους για την οικονομία, βλέπουμε ότι χρειάζεται η Ευρωστάτ να έχει τους απαραίτητους πόρους ούτως ώστε να έχει και τις καλές στατιστικές και να μπορέσει να χρησιμοποιεί τι θετικέ που έχει. Αλλιώ θα έχουμε προβλήματα. Ελπίζω λοιπόν να γυρίσουμε, συνεχίσουμε προ την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, εγώ σα ευχαριστώ. Θέλει κανένα άλλο το λόγο για το θέμα αυτό. Όχι. Κύριε Λούφιξον, μήπως θέλετε να απαντήσετε σε κάτι. Jag tackar för diskussionen och Μου φαίνεται ότι συμφωνούμε. Συμφωνούμε για τα διάφορα σημεία που έθιξα και στα γενικά μας συμπεράσματα. Να προσθέσω ότι μπορεί να μας φαίνεται ότι έχουμε πολύ χρόνο στο τέλος Αυγούστου, ωστόσο θα είμαστε σε διακοπές όταν θα πρέπει να λάβουμε θέση σε σχέση με τις τροπολογίες. Εάν λοιπόν έχετε κάτι να επισημάνετε σε σχέση με τις τροπολογίες, θα ήθελα να τις λάβω στα δυνατόν συντομότερα για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε, να καταλήξουμε στην τελική μας απόφαση ήδη από το τέλος Αυγούστου. Σας ευχαριστούμε. Φέρετε ότι το χρονοδιάγραμμα εδώ είναι κάπως παράξενο πρόκειται να σας απασχολήσει και στις διακοπές σας. Η υποβολή για, την, για τις τροπολογίες, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 20 Ιουλίου, αλλά υπάρχει και άλλη προθεσμία για τις τροπολογίες σε σχέση με τον προπολογισμό που αφορούν το άλλο έγγραφο. Εκεί 19 Αυγούστου είναι τροπολογία. Αυτό μου λένε μετά θα ψηφίσουμε την έκθεση 31 Αυγούστου και ψηφοφορία στην Επιτροπή θα έχουμε τον Οκτώβριο, ώστε να περάσει και στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Ελπίζουμε να προλάβουμε με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Αν κανεί θέλει κάποια διευκρίνηση και τι σημαίνουν όλα αυτά, ελάτε σε επαφή με τη Γραμματεία, εάν έχετε την παραμικρή αμφιβολία σε σχέση με τι δημοσιονομικέ, όπω ονομάστηκαν, τροπολογίε. Και τώρα να περάσουμε στο σημείο 13 τη ημερήσια διάταξη για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση στην εσωτερική αγορά. Έκθεση τη κυρία Οκονή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με δύο λόγια θα σας παρουσιάσω το περιεχόμενο. Το 2009 το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό, δηλαδή τα τυχερά παιχνίδια ε, online, σε απευθεία σύνδεση, μετά από μια συναδέλφου που Κριστέλ Σαλντομόζ. Ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τις οικονομικές και μη οικονομικές επιπτώσεις ε, για τη διασυνοριακή ε, προσφορά υπηρεσιών. Η Επιτροπή πέρυσι ε, το Μάρτιο παρουσίασε μια πράσινη βίβλο που αρχίζει να καθορίζει για το θέμα αυτό το αν πρέπει να αφήσουμε ελεύθερα τα κάτι μέλη με τις διαφορές τις οποίες έχουν ή αν πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή κάποια ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά από τον τελευταίο Μάρτιο. Να σας δώσω και κάποια αριθμητικά στοιχεία που είναι σημαντικά για να παρουσιάσουμε την οικονομική βαρύτητα του τομέα. Δεν είναι αμεληταίος. Τα αιτήσια έσοδα στην Ευρώπη ξεπερνάνε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008. Η Ευρώπη ε, έχει 45, αποτελεί το 45% της παγκόσμιας αγοράς. Ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών αποτελεί 7,5% διορθώνει ομιλείται το, ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί το 7,5% ε, του τομέα των τυχερών παιχνιδιών γενικότερα που μέχρι το 2013 φαντάζομαι ότι θα διπλασιαστεί αυτό το, ποσοστό. Σα τα λέω για να σα παρουσιάσω τη βαρύτητα του τομέα. Δεν είναι καθόλου αμεληταίος ε, και έχει και ταχύτατη ανάπτυξη. Το οικονομικό δυναμικό του τομέα έχει καταστεί σαφές ε, σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να το εκμεταλλευτούν και επειδή υπάρχει ε, μεγάλη διαφορά στις ε, εθνικές διατάξεις και υπάρχει και μεγάλη ποικιλία εμπλεκομένων έχουν, έχει δημιουργηθεί, έχει δημιουργηθεί μια παράνομη αγορά και είναι και ένα τομέα εύκολου ξεπλήματο χρήματο. Γι' αυτό είναι προ συμφέρον μας ε, να αποτρέψουμε τους παίκτες από ε, τις παράνομες προσφορές τυχερών παιχνιδιών. Αυτό είναι προ όφελό μας και είναι και ε, υπέρ των νόμιμων φορέων στοιχηματισμού και τυχερών παιχνιδιών. Τα παράνομα παιχνίδια οδηγούν σε προσπάθειε ε, χειραγώγησης των αποτελεσμάτων και ο αθλητισμός είναι ευάλωτο σε τέτοιες απειλέ, γιατί αυτές οι απειλέ ε, ε, αφορούν και τα γνωστά αθλήματα αλλά και πολλές φορές και αγώνες μικρότερη σημασίας ή αθλήματα μικρότερη σημασία. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας διότι κατά αυτό τον τρόπο οδηγούμεθα σε μια διαφορία για τον αθλητισμό. Ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιστεύω ότι πρέπει πρώτον να εγγυηθούμε την προσφορά της νόμιμης ε, ε, των νόμιμων υπηρεσιών Δεύτερον, θα πρέπει να εγγυηθούμε μια συνεχή οικονομική σχέση μεταξύ των εσόδων από τα αθλητικά στοιχήματα και των αθλητικών διοργανώσεων και αυτή η πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει να κατευθυνθεί προς την προστασία των αγωνισμάτων κατά της απάτης και υπέρ της ε, μαζικής ανάπτυξης του αθλητισμού. Τέλος, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μείζωνα ευθύνη για την προστασία της ακαιρεότητας του αθλητισμού και ευχαριστώ πολύ τον Ζων Πολ που έχει μείνει ως εδώ για να με παρακολουθεί γιατί δεν είναι και πολλοί συνάδελφοι και συνοψίζω ε, λέγοντας ε, ότι προτείνω να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός ε, ένας οργανισμός, φορέας, δεν ξέρω πώς θα τον πούμε, για την ακαιρεότητα του αθλητισμού με βάση το άρθρο 6, 83 και 155 της συνθήκης για την προώθηση της εκπαίδευσης ε, και των νέων και των αθλητών για την αποφυγή της διαφθοράς στον αθλητισμό βελτιώνοντας ε, την πληροφόρηση και βασιζόμενη σε ένα κοινό σύστημα αξιολόγηση των παραβάσεων και κυρώσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για, την, την, παρουσία σας εδώ και για την προσοχή σας. Yes, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ομιλητές έχουν ζητήσει το λόγο. Ντέρκ πρώτα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πράσινη βίβλα σε Επιτροπή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Η Κομισιόν διατυπώνει όμως τα κείμενά της με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν ξέρει πολλά πράγματα για το θέμα αυτό. Είναι ανοιχτά τα ερωτήματα της Κομισιόν κατά βάση. Μας δίνει μόνο κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρει πολλά πράγματα. όσον αφορά αυτά που αναφέρονται στην Πράσινη Βίλβο σημαίνουν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ελέγξουν αυτές τις διαστηριότητε στις χώρες τους καλώς και θα πρέπει να εξεταστεί επίσης κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να προσφέρει προστιθέμενη αξία όσον αφορά αυτά τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Θα δούμε κατά πόσον είναι καλό να έχουμε συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών γιατί αυτό το φαινόμενο δεν περιορίζεται από τα σύνορα μιας χώρας. Ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εδώ για υπηρεσία η οποία εξαιρείται το από την οδηγία ε, τέλος πάντων περίεργο που έχουμε εδώ μια εξαίρεση τι να κάνουμε αλλά πρόκειται για μια υπηρεσία, προσφορά μιας υπηρεσίας και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους και πώς και κατά πόσον η Κομισιόν δεν θα μπορούσε να είναι πιο συντομισμένη. Έχει δίκιο η συνάδελφο ότι υπάρχει έντονο οικονομικό συμφέρον των ε, δραστηριοτήτων αυτών και αρκετά σημαντικό. Το φαινόμενο αυτό ξεπερνά τα σύνορα, άρα χρειάζεται συντονισμό. Και επαναλαμβάνω ότι πρέπει οπωσδήποτε να απαγορεύσουμε και να καταπολεμήσουμε όλα τα παράνομα ε, παιχνίδια. Τώρα κατά πόσο η αγορά αυτή είναι μαύρη, μονοφαιά θα το δούμε. Αλλά το θέμα της εγκληματικότητας ε, είναι πάρα πολύ πραγματικά επικίνδυνο. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε και να καταλήξουμε σε κάποιους διακανονισμούς. Είναι καλύτερο να έχουμε ένα πλαίσιο για νο... νόμιμα παιχνίδια άμεση σύνδεση. Πιο καλά παρά να τα αφήσουμε έτσι παράνομα. Είναι σαν να λέμε ότι απαγορεύεται Και βλέπουμε όμως καμιά φορά τι γίνεται στην Κίνα. Εντάξει, τα πράγματα είναι περίεργα εκεί. Ε, να πούμε, σαν να λέμε απαγορεύεται το κάπνισμα, αλλά κάπου πρέπει κάποιος να καπνίζει και νόμιμα. Και κυρίως θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Οι εν λόγω επιχειρήσει θα πρέπει να έχουν και την σωστή οικονομική συμπεριφορά. Είναι σωστό πολλές από τις παρατηρήσεις της Σοκουνή που αναφέρθηκε στον αθλητισμό και αναφέρθηκε στα παράνομα στοιχήματα και όλα αυτά θα πρέπει να διεξετάσουμε. Νομίζω ότι έχουμε παραβλέψει ίσως αυτό το συσχετισμό ανάμεσα στα στοιχήματα και στον αθλητισμό. Από την άλλη μεριά Πολλέ από τις διασυνδέσεις αυτές ίσω είναι θετικέ. γιατί πολλά από τα έσοδα είναι προ όφελο του αθλητισμού του ίδιου. Εμείς ε, δεν θα πρέπει εδώ να παραμείνουμε προσκολλημένοι στον αθλητισμό αλλά να ζητήσουμε γενικό διακανονισμό, διαφάνεια και νόμιμα παιχνίδια επίσης. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν πιο ανοιχτή αλλά πιο κλειστή πολιτική στοιχημάτων. Εκείνοι που είναι πιο κλειστοί βέβαια πιέζονται από τα άλλα κράτη-μέλη και δεν είναι το καλύτερο να παρέμβει η Ευρώπη θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη απλώς να συντονιστούν. Θα αρκούσε μου φαίνεται. Δεν θέλουμε μια νέα υπηρεσία. Καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών. Ευχαριστώ. Uh, ένα σημείο κίνηση είναι ότι δεν υπάρχει νομοθετικό εναρμοσμένο πλαίσιο, άρα η ελευθερία εγκατάσταση και η ελευθερία προσφοράς υπηρεσιών είναι αυτές που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Στην πραγματικότητα, ο νέας αυτός των παιχνιδιών βρίσκεται ένα κατακαιρματισμό των ε, αγορών με τους ε, ενδιαφερόμενους να βλέπουν να υπάρχουν προβλήματα μια χώρα στην άλλη. Οι εθνικέ άδειες θα πρέπει λοιπόν να είναι εξαίρεση όσον αφορά τις λειτουργίες αυτές και να μην επιβάλλουν σαν κανόνας. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μια καθαρά εθνική πολιτική. Προκειμένου να δικαιολογηθεί η παραγωγή και να συμμορφωθούμε με τις αρχές που ορίζει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ιδίως σε σχέση με την αναλογικότητα των μέτρων περιορισμού. Σε συμπέρασμα, να εκφράσω το, ότι χαιρετίζω τη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα αμοιβέ αναγνώριση μεταξύ των φορέων των κρατών μελών που έχουν εγκριθεί. Και αυτό για να υπάρξει υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών και τη δημόσια ε, τάξη. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Ο κ. Χουντή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ζητώ συγγνώμη διότι δεν μπόρεσα να ακούσω την εισήγηση της συναδέλφου η κατάσταση στην Ελλάδα μας έχει σωμηρία με τα κινητά και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν την άκουσα την εισήγησή σας. Παρ' όλα αυτά έχω διαβάσει τη γνωμάτευση, τη γνωμοδότηση. Έχω την εντύπωση παρά τη φιλότιμη προσπάθεια, είναι άτολμο το κείμενο, όπως είναι, άτολμη και, είναι και η έκθεση η, της αρμόδιας επιτροπής. Τι θέλω να πω με αυτό. Το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο από ό,τι το αντιλαμβανόμαστε. Είναι δύσκολο να συνδυάσεις το παιχνίδι, το τζόγο, με την προστασία του αθλητισμού και την προστασία του πολίτη. Η εμπειρία μου πλούσια προέρχεται κυρίως από το χώρο του ποδοσφαίρου. Αλλά και γενικότερα νομίζω ισχύουν όλα αυτά που θα προσπαθήσω να σας πω ο τζόγος, ο ανεξέλεκτος, δημιουργεί και αλλοιώνει και τα αποτελέσματα τα αθλητικά, με συνέπεια να έχουμε έντονα φαινόμενα διαφθοράς, διαπλοκής, ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε απερίγραπτες διαστάσεις. Τι να σας πω. Ξεπερνάνε και εθνικούς προϋπολογισμούς. Και αποτελούν και καταστροφή για τα αθλήματα και για τον αθλητισμό παραδείγματος χάρη λέγεται κάπου ότι αυτή η δραστηριότητα φέρνει χρήματα και χρηματοδοτεί τον αθλητισμό. Αυτό εν μέρει είναι σωστό. Διότι η πρώτη λειτουργία, η αλλίωση των αποτελεσμάτων, αυτός ο ανεξέλεκτος τζόγος διώχνει τον κόσμο από τον αθλητισμό. Διώχνει τους φιλάθρους από τις κερκίδες διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι παρακολουθούν ένα τίμιο αγώνα. Και επομένως η οικονομική αναπλήρωση δεν λύνει το πρόβλημα, μάλλον το διονύζει και θεωρείται ότι είναι η λύση του προβλήματος. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα της προστασίας των ανηλίκων κτλ. Τώρα, ε, στις προτάσεις. Δεν μπορεί να μένουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης απλώς στις αρχές που λέει η συνθήκη στο 165 και ούτω καθεξής. Υπάρχουν τρόποι και τεχνικές που μπορεί να συμμαζευτεί λίγο το πράγμα και μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μπορεί και να ελεγχθεί και να υπάρξει ένας μηχανισμός πρόληψης εκεί που πάμε να ξεφύγει όλη αυτή η κατάσταση η οποία είναι δύσκολη το παραδέχομαι να συμβιβάσεις το δικαίωμα ο άλλος να τζογάρει online, να παίζει προσδοκώντας υψηλά κέρδη και ταυτόχρονα αυτό να είναι υπέρ της προστασίας του αθλητισμού. Δυστυχώς στις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς και των υπηρεσιών που ζούμε <laughs> δεν μπορεί να πας σε μεγαλύτερες απαγορεύσεις και το βλέπω. Αν και όταν τα απαγορεύεις ορισμένα πράγματα το παράνομο βρίσκει εύκολο τρόπο και επιδεινώνεται παραδέχομαι η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει είναι μια βάση το σχέδιο για να τελειώσω. Το θεωρώ άτολμο. Θα συνεργαστούμε με την εισηγήτρια από την οποία ζητώ συγγνώμη αν κάποια θέματα που έθιξα τα είπε στην εισήγησή της, να το κάνουμε καλύτερο, να βοηθήσουμε να γίνει, αν είναι δυνατόν, καλύτερο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Σοφή, εάν θέλεις να επανέλθεις, σύντομα, γιατί θα φύγουν οι διερμηνείς. Φαντάζομαι ότι έχεις λίγες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημειώνω τις παρατηρήσεις, τα σχόλια των συναδέλφων. Απλώς, για όσοι από κύριο Στέξ που δεν είναι εδώ, να του πω ότι δεν θέλω να κοντράρω τα στοιχήματα ή τα τυχερά παιχνίδια ακριβώς. Όχι, υπάρχουν και οικονομικά διακυβέρματα που θα μπορούσε να προκαλούν και φαινόμενα διαφθορά ή απάτης. Εκεί θα πρέπει να δείξουμε όλοι μας την επαγρύπνηση και δεν λέω απλώς ότι δεν πρέπει να αντιτιθέμεθα, αλλά μάλιστα να συμμετάσχουμε στην εξέλιξη, τη χρηματοδότηση του αθλητισμού μαζικά, εάν γίνεται, χάρη στα κέρδη που μπορούμε να αποσπάσουμε από τα παιχνίδια στο διαδίκτυο. Είναι σημαντική πηγή εσόδων. Τώρα, ω προ τι φιλοδοξίε του κειμένου η κατάσταση σε κάθε κράτος το πώς είναι τα τυχερά παίγνια ειδικά στο διαδίκτυο είναι κάτι που την χάνει διαφορετικής προσέγγισης. Είναι δύσκολο σήμερα, ακριβώ επειδή υπάρχουν τόσες διαφορές μεταξύ κρατών, να έχουμε ένα υπερφιλόδοξο κείμενο ώστε να υπάρξει και εναρμόνιση. Εδώ έχουμε ένα μόνο πρώτο, πρώτο βήμα. Ελπίζουμε ότι στο χρόνο θα μας επιτρέψει να έχουμε καλύτερες εξελίξεις και ευχαρίστως να ακούσω τις δικές σας τις ερμηνείες και τα σχόλια για να βελτιώσω το δυνατόν το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 15 Ιουλίου, εξέταση 31 Αυγούστου και ψηφοφορία πάλι στις 31 Αυγούστου. Στην ΙΜΚΟ 19 Σεπτεμβρίου με στόχο να περάσει στη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου η έκθεση. Ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν διάφορα. Η ημερομηνία της προσεχούς συνεδρίασης Τετάρτη 31 Αυγούστου στις 9 το πρωί. Και πάλι το απόγευμα στις 3. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Γεια σας.